Uh, Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε μάλλον αυτή την ακρόαση σχετικά με τις γυναίκες και την κλιματική αλλαγή. Θα συνεχίσω στη γλώσσα μου, γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ τα ακουστικά σας. Λοιπόν, έχουμε αυτή την ακρόαση και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία τα σχόλια της παρεμβάσης ε, των εμπειρογνωμόνων. Το θέμα του κλίματος είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους και η παρούσα και μελλοντική κλιματική αλλαγή οπωσδήποτε θα έχει επιπτώσεις σε όλους μας. Βεβαίω, καταλαβαίνετε ε, και είναι σαφές ε, ότι η κλιματική αλλαγή δεν έχει ίδια επίπτωση σε όλους. Πλήττει πολύ περισσότερο το νότιο ημισφαίριο και τους φτωχούς ε, λαούς, πολύ περισσότερο λέω από ότι ε, τις χώρες του Βορρά. Επίσης οι γυναίκες πλήγονται περισσότερο από τους άντρες. Γι' αυτό ακριβώς επιλέξαμε σαν θέμα της σημερινής ακροάσεως ε, το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τις γυναίκες είναι σημαντικό να έχουμε εργαλεία, να έχουμε δυνατότητες επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με το ζήτημα αυτό έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το μέλλον, να δούμε είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Ε, ξέρουμε ότι ε, τώρα στη σύγχρονη κοινωνία παίρνουμε συνέχεια το αυτοκίνητό μας, ε, καταναλώνουμε βενζίνες, καταστρέφουμε το περιβάλλον, κάνουμε πολλά πράγματα τα οποία είναι κακά και άσχημα. Για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε και κάτι καλό ε, λοιπόν, ε, θα έχουμε, έχουμε και την ε, Επίτροπο κυρία Κόνι Χέντεγκάρντ, η οποία κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. θα δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα στην Νικόλ Κιλ και μετά στην Επίτροπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν αναφερθώ συγκεκριμένα στην ε, στο θέμα μας. Θα ήθελα να έχουμε μία σκέψη για την Ουάγκαρη Ματάη που μας εγκατέλειψε πρόσφατα, μας άφησε πρόσφατα. Να θυμίσουμε μια φράση της ε, που είναι πολύ εύγλωτη ε, είναι φράση της συζύγου, του συζύγου συγγνώμη, που ζητώντας το διαζύγιο είπε είναι υπερβολικά λαμπερό μυαλό, υπερβολικά ε, ε, ε πισματάρα, ε, υπερβολικά δύσκολο να την ελέγξει κανείς. Έχει μεγάλη εκπαίδευση και είναι και πολύ έξυπνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν μιλάμε για τη γυναίκα η οποία δημιούργησε την ιδέα και το κίνημα της πράσινης ζώνης. 47 εκατομμύρια ε, δέντρα και ε, χιλιάδες θέσεις εργασίας για τις γυναίκες γιατί η Όγκαρη ήταν πολύ δεσμευμένη και στρατευμένη στο θέμα των γυναικών έδωσε επίσης την ε, δυνατότητα να αλλάξει η εικόνα της γυναίκας στην Αφρική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Να αποκτήσει αξία η εικόνα της Αφρικανής γυναίκας που δεν θα έπρεπε πλέον να τη βλέπουμε σαν θύμα αλλά και σαν ε, ένα ανθρώπινο όνο το οποίο μπορεί να ελέγξει το, τη μοίρα του. Επίσης να θυμίσουμε και την φράση στην οποία βασίστηκε η Επιτροπή που της απένουμε το βραβείο Νόμπελ βάσει του βραβείου ε, θελήσαμε να επιβραβέσουμε τη στάση της όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως δε των προβλημάτων των γυναικών ε, και την αξιοποίηση της ε, γυναίκας για σκοπούς ειρήνης και ανάπτυξης. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής ε, γιατί σήμερα έχουμε εδώ τόσο διαφορετικούς εμπειρογνώμονες που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ε, δούμε τις διάφορες πλευρές αυτού του περίπλοκου και πλούσιου ζητήματος. Θέμα μας λοιπόν είναι οι κλιματικές αλλαγές και οι γυναίκες. Ε, και ξέρετε, εγώ πρέπει να κάνω και έκθεση για το θέμα αυτό. Και όταν λέω θέλω, πρέπει να δουλέψω για το θέμα κλιματικές αλλαγές και γυναίκα, δεν καταλαβαίνουμε και πάρα πολύ καλά περί τίνο πρόκειται. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα το οποίο εμπνέει πολύ τον κόσμο γιατί θέλουμε ας πούμε, να ξεχωρίσουμε τις γυναίκες απέναντι στην κλιματική αλλαγή, μια και άνδρες και γυναίκες υποτίθεται ότι ζούμε μαζί στον ίδιο πλανήτη. Μα γιατί πιστεύουμε ότι οι κλιματικές αλλαγές δεν θα ε, έχουν τον ίδιο αντίκτυπο ε, σε όλους. Υπάρχουν ε, κάποια νησιά του Ειρηνικού που κινδυνεύουν μετά από 50 χρόνια να εξαφανιστούν. Ενώ ας πούμε σε μια πλούσια γειτονιά Στι στις Ηνωμένε Πολιτείε, στη Νέα Υόρκη, ενδεχομένως δεν θα καταλάβουν και πολλά οι κάτοικοι από τις κλιματικές αλλαγές. Επομένως και η πολιτική σταθερότητα ε, και οι παραδοσιακές δομές αλληλεγγύης και οι θεσμικά ε, κατοχυρωμένες κοινωνίες ε, θα κρίνουν την ικανότητα και την δυνατότητα που θα έχει το κάθε άτομο να ξανασταθεί στα πόδια του. Πού βρίσκονται οι γυναίκες ε, μέσα σε όλο αυτό το θέμα, θα με ρωτήσετε. Δεν θα έπρεπε καλύτερα να θέσουμε διαφορετικά το ερώτημα, να έχουμε ένα θέμα ας πούμε φτώχεια, ένδια και κλιματική αλλαγή, επαγγελματική αστάθεια και κλιματική αλλαγή. Σας απαντώ όχι, γιατί ε, δεν υπάρχει ομοιογένεια σε όλο τον πλανήτη, δηλαδή δεν έχουν όλα τα ίδια χαρακτηριστικά σε ολόκληρο τον πλανήτη, ούτε καν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βεβαίως Α, συγγνώμη, διορθώνει η ομιλήτρια. Βρίσκουμε, βρίσκουμε κοινά χαρακτηριστικά, διορθώνει η ομιλήτρια, ε, σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολύ κοινά χαρακτηριστικά για τις γυναίκες ε, η εγκυμοσύνη, ο τοκετός, η δυνατότητα διαχείρισης ε, του αναπαραγωγικού δικαιώματός τους, η μηνιαία έμεινος ρίση, όλα αυτά είναι κοινά Επίσης, οι γυναίκες ενώ οι αντιπροσωπεύουν το 70% των ανθρώπων που ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο τη μέρα έχουν λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας ιδιοκτησίας. Επίσης αντιπροσωπεύονται ε, στις θέσεις εξουσίας και λήψης απόφασης. Έχουμε 17% γυναίκες βουλευτές ε, στον όλο τον κόσμο και 8% γυναίκες υπουργοί. Είναι γεγονός ότι στη Δανία έχουν γίνει γίνει πολλές προσπάθειες έτσι ώστε να ανεβεί ο μέσος όρος των στατιστικών. Οι γυναίκες λοιπόν είναι αυτές οι οποίες δουλεύουν ε, περισσότερο με μη αμοιβόμενη εργασία παρέχοντας ε, βοήθεια και ε, και φροντίδα σε παιδιά, σε ηλικιωμένους, σε ανάπηρους και επομένως είναι οι γυναίκες οι οποίες στο μέγιστο βαθμό συμβάλλουν στην παγκόσμια εργασία αλλά μονάχα με 10% της παγκόσμιας παραγωγής χρήματος και βεβαίως οι γυναίκες είναι τα πρώτα και μεγαλύτερα θύματα του εμπορίου ανθρωπίνων όντων ε, και οι γυναίκες, δεν πρέπει να ξεχνούμε, αντιπροσωπεύουν το 80% των εκτοπισμένων και των προσφύγων. Ορίστε, μία σειρά στοιχείων που καταδεικνύουν ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να ε, βάλουμε τις γυναίκες σαν ένα ηλαιό ε, της αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών. Φτάνει και η Επίτροπος και επομένως είναι πάρα πολύ καλό, θα μπορούσαμε να του δώσουμε και το λόγο. lui donner la parole, on est d'accord. Ja, jag är glad att vi nu har fått... Πολύ ωραία. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε πλέον την ε, Επίτροπο ε, μαζί μας, την κυρία Κόνη Χέντεγκαρντ, η οποία είναι Επίτροπος υπεύθυνη για το κλίμα. Και θα της δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι διότι με καλέσατε εδώ και Είχα την ευκαιρία να διαβάσω και τις προηγούμενες παρουσιάσεις. Επομένως, ε, έχω ενημερωθεί κάπως για τις εξελίξεις στη δική σας Επιτροπή. Ξέρουμε ότι η κλιματική αλλαγή απειλεί να διαβρώσει την, την ε, ανθρώπινη ελευθερία. Θα οδηγήσει σε περισσότερες ανισότητες σε όλα τα επίπεδα. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει διαφορετικά τους άνδρες και διαφορετικά τις γυναίκες. Διότι ε, ε, ε, επισέρχονται όχι μόνο οι περιβαλλοντικές συνθήκες αλλά και οι κοινωνικές συνθήκες. Ο αναπτυσσόμενος κόσμος θα επομιστεί μεγαλύτερο βάρος και οι γυναίκες στις πιο φτωχές και στις, πιο στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι αυτές που θα πληγούν περισσότερο. Το 70% ε, των ε, ανθρώπων που ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα είναι γυναίκες. Ε, έχουν καθεστώς περιθροποίησης και έτσι φέρουν δυσβάσταχτο και δυσανάλογο βάρος. Στον Μπαγκλαντές, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, στον Μπαγκλαντές μετά από την έλευση ενός πολύ μεγάλου τυφώνα η αναλογία γυναικών θυμάτων ήταν πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή πέντε γυναίκες θύματα προς ένα άνδρα. Και έτσι αυτό οφειλόταν σε, και σε πολιτιστικές αλλαγές. Δηλαδή ότι η γυναίκα δεν είχε το δικαίωμα να φύγει από το σπίτι της χωρίς να συνοδεύεται από ένα άνδρα. Άρα αναγκάστηκε να μείνει με στο σπίτι όταν ήδη ερχόταν η πλημμύρα. Ήταν αιτία για την κατάσταση αυτή. Πρόσβαση στην ενέργεια επίσης. Αν ε, πρέπει κανείς να πάει πάρα πολύ μακριά για να βρει ξύλα να ανάψει τη φωτιά στο σπίτι, τότε η πιθανότητα ε, το κορίτσι αυτό να πάει στο σχολείο μειώνεται δραστικά γιατί οφείλει να ε, κάνει όλο και μεγαλύτερη απόσταση για να βρει ξύλα να τα βάλει στη φωτιά στο σπιτικό και γι' αυτό λέμε ότι οι κλιματολογικές αλλαγές πλήττουν τις γυναίκες περισσότερο. Οι γυναίκες και οι άνδρες σίγουρα δεν εκτίθενται επίσης όρις στις κλιματικές αλλαγές και δεν έχουν και τις ίδιες προσαρμοστικές δυνατότητες λόγω των ανισοτήτων σε οικονομικό και κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Αλλά και η μετανάστευση πλήττει τις γυναίκες με διαφορετικό τρόπο οι γυναίκες που μεταναστεύουν διακινδυνεύουν περισσότερο να εκτεθούν σε βία βασισμένη στη διάκριση των φύλων. Η επανεγκατάσταση επλήττει ιδιαίτερο στα δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης. Οι φτωχές γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε φυσικούς όρους, ε, πόρους, στην τεχνολογία και σε διάφορα άλλα μέσα και επομένως δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις φυσικές καταστροφές. Παραδοσιακά οι διαφορά μεταξύ των δύο ρόλων οξύνεται και μειώνεται η πιθανότητα τα νεαρά κορίτσια να μπορέσουν να διαφοροποιήσουν το ε, πεπρωμένο τους. Θα πρέπει λοιπόν να τις αναγνωρίσουμε αυτές τις ε, διαφορές και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου τα μέτρα προσαρμογής να έχουν επιτυχία. Οι γυναίκε είναι καθοριστικός παράγοντας για να προσαρμοστεί η καθημερινότητα στην κλιματική αλλαγή. Χρειαζόμαστε τη γνώση των τοπικών συνθήκων. Για παράδειγμα, οι γυναίκες που ανήκουν σε φυλές Ινδιάνων, οι θαγενεί ε, ε, κάνουν διάφορες δράσει επαναφύτευση στα μέρη όπου ζουν όσοι λαμβάνουν μέρο στη διαδικασία λήψη αποφάσεων θα πρέπει να αφουγκραστούν αυτές τις γυναίκε και να χρησιμοποιήσουν όλη αυτή τη ε, γνώση στην προσπάθεια μετριασμού ε, των ε, περιβαλλοντικών προβλημάτων. Από εκεί και πέρα οφείλουμε επίσης να λάβουμε υπόψη μας πολλά άλλα θέματα όπως είναι η πρόσβαση των γυναικών στους φυσικούς πόρους και στον έλεγχο αυτό αυτών. Να αξιοποιήσουμε καλύτερα τη γνώση τους για να μετριάσουμε τις καταστροφές και να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να βελτιώσουμε την πρόσβαση των γυναικών στην πληροφόρηση, στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για τις καταστροφές, ε, στα συστήματα ενημέρωσης για τις αλλαγές του καιρού. Οι γυναίκες που δεν έχουν ε, επαρκές εκπαιδευτικό επίπεδο δεν θα πρέπει για το λόγο αυτό να αποκλείονται από την ενημέρωση και την πληροφόρηση. Πολύ συχνά παραγνωρίζεται η διάσταση του φύλου στη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή. Οι ομάδες που εκπροσωπούν οργανώ, γυναικείς οργανώσεις, οι ομάδες που εκπροσωπούν τις γυναίκες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι παράγοντες θα πρέπει να ασκήσουν περισσότερη πίεση ώστε η στρατηγική για το 2020 που θα αφορά τόσο τις ε, βιομηχανικές χώρες όσο και τις αναπτυσσόμενες να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τη διάσταση του φύλου. Βεβαίως θα βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή και τις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μέσα στις χώρες αυτές, όπως είναι οι γυναίκες και τα παιδιά. Θα έχουμε μια προσέγγιση twin track σε διπλό δρόμο και θα σας δείξω ορισμένα παραδείγματα. Για παράδειγμα στη Βραζιλία, τι ακριβώς κάνουμε. Διευκολύνουμε τις γυναίκες να βρουν θέσεις απασχόλησης, καλλιεργώντας ε, ε, βιώσιμες καλλιέργειες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για βιώσιμη παραγωγή και αηφόρο παραγωγή καυσίμων. Πολλές δράσεις μπορούν να γίνουν και γίνονται. Εν συντομία όμως, θα ήθελα να πω το εξής. Ναι, ε, έχουμε καλά παραδείγματα τα οποία, στα οποία κάνουμε mainstreaming και τα βάζουμε στο επίκεντρο της ε, ατζέντα μας, ωστόσο πρέπει να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας. Στα αναπτυξιακά προγράμματα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη διάσταση του, του φύλου. Είναι κάτι το σχετικά καινούριο αυτό το σκεπτικό. Όλα τα προγράμματα ε, που έχουν σχέση με το κλίμα θα πρέπει να τα εξετάσουμε προσεκτικά και να δούμε κατά πόσο ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου. Δηλαδή, τη γενική στρατηγική την έχουμε, στην εφαρμογή όμως και στην υλοποίηση πρέπει να εξετάσουμε πιο προσεκτικά το τι ακριβώς συμβαίνει. Τέλος, θα ήθελα να πω και το εξής. Στη διάσκεψη για το κλίμα στην Κανκούν, για πρώτη φορά έγινε λόγος για τη διάσταση ε, του φύλου. Αναγνωρίστηκε ότι τα θέματα που αφορούν τις γυναίκες, την ισότητα των δύο φύλων, είναι απαραίτητο να ενσωματώνονται στον αγώνα για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Και στα επικουρικά σώματα επίσης υιοθετήθηκε αντίστοιχη διατύπωση αλλά και στην εθνική εφαρμογή των εκάστοτε σχεδίων ε, θα πρέπει να υιοθετηθεί αντίστοιχη διατύπωση Και θα ήθελα να πω επίσης ότι με η κοδεσπότη την Πατρίσια Εσπινόσα είχαμε μια συνάντηση Τρόικας με παρόντες εκπροσώπους της κυβερνήσης της Δανίας, της Νότιου Αφρικής και του ε, Μεξικό και έγινε προετοιμασία εν ώψη της επόμενης συνάντησης στον, Durban. Θα συνεργαστεί επίσης η Κριστιάνα Φιγκέρες από το UNFCC και η Μέρι Ρόμπινσον που γνωρίζετε πολύ καλά όλοι. Είναι, είμαι πολύ περήφανη που θα συνεργαστώ με αυτή την ε, ομάδα και σε όλες τις διασκέψεις για το κλίμα θα, θα γίνει δουλειά ώστε να συμπεριληφθεί ε, πιο ενεργά η διάσταση του φύλου. Νομίζω ότι η κυβέρνηση της ε, της Νοτιού Αφρικής, η οποία θα φιλοξενήσει το COP17, έχει προγραμματίσει διάφορες δραστηριότητες. και θα γίνει και ε, συνάντηση της ομάδας υψηλού επίπεδου για τα θέματα των γυναικών. Και εκεί θα παραστούν πολλές γυναίκες υπουργοί και ελπίζουμε και άνδρες υπουργοί, έτσι ώστε όταν ε, συζητήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα, με όλο το σεβασμό που σας τρέφω, να μην καταλήξει να είναι μια συνεδρίαση ε, στην οποία θα παρίστανται ένα σωρό γυναίκες. Θα πρέπει να είναι μια γενική συνεδρίαση στην οποία να παρίστανται όλοι για να, για να αποδείξουμε στην πράξη το mainstreaming, το ότι δηλαδή τα θέματα της ισότητας των φύλων βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής μας. Είναι πολύ καλή αυτή η πρωτοβουλία γιατί πρέπει να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας ε, στον τομέα της εφαρμογής της γενικότερης στρατηγικής μας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις. Σας είμαστε ευγνώμονες διότι πραγματικά βρήκατε χρόνο στο πρόγραμμά σας να έρθετε να μας δείτε, να μας μιλήσετε και νομίζω ότι παρουσιάσατε πολύ καλά παραδείγματα για το τι γίνεται με την ισότητα των φύλων και τις κλιματικές αλλαγές. Βεβαίως θα επανέλθουμε σε όλα αυτά τα ζητήματα και θα ήθελα αυτή τη στιγμή να σας παρουσιάσω δύο εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα μιλήσουν 15, από 15 λεπτά ο καθένας. Έχουμε την Ιρένε Ντάνκενμαν από το Πανεπιστήμιο του Μαντχέιμενγκεν. Ιρένε, έχετε το λόγο. Thank you very much and... Ευχαριστώ. Χαίρομαι που βλέπω τόσα πολλά πρόσωπα εδώ μέσα στην αίθουσα. Δείχνει αυτό ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα που συζητούμε. Εγώ είμαι τεχνική ε, ως, ε, έχω σπουδάσει τεχνική, ένα τεχνικό επάγγελμα, οικολογία και έχω δει πώς ακριβώς ε, σχετίζεται αυτό με την κοινωνική διάσταση. Έχω δουλέψει με ομάδες γυναικών και αντρών σε όλο τον ε, κόσμο και γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι το θέμα του φύλου. Η δική μου παρουσίαση έχει να κάνει με το να δώσουμε ένα ανθρώπινο πρόσωπο σε αυτό το θέμα. Θα μιλήσω τη μετρική μου, Ολλανδικά δηλαδή. Ελπίζω να μπορέσετε να παρακολουθήσετε και το πάθος που έχω για το θέμα αυτό. Δεν έχω δυστυχώς παρουσίαση PowerPoint, μόνο κάποιες, ε, με κείμενο, μόνο κάποιες ε, εικόνες θα μπορώ να σας δείξω. Οι κλιματικές αλλαγές συχνά παρουσιάζονται ως ε, τεχνικό και πολιτικό θέμα, το οποίο προκύπτει σε διεθνές επίπεδο. Ξεχνάμε όμως ότι ε, ποια είναι η ανθρώπινη πτυχή στις κλιματικές αλλαγές. Οι άνθρωποι και η συνύπαρξή τους είναι, σημαντικό, είναι σημαντική πτυχή και θα πρέπει να το δούμε σε σχέση και με τις κλιματικές αλλαγές. Πρέπει να δούμε πού μπορούμε να ε, προσφέρουμε έτσι ώστε να, υπάρχει, να μειωθούν οι φιλετικές και οι κοινωνικές ανισότητες. Η κυρία Ατίμψελ Αμπάντε από την Κάνα είναι 45 χρονών, τη βλέπετε, και λέει ότι έχω 7 παιδιά, ε, το σπίτι μας καταστράφηκε μετά από μία πλημμύρα και ε, τα σιτηρά που είχαμε απλώς ε, τα πήρε το ρεύμα. Και τώρα πραγματικά υποφέρουμε από την πείνα για πολλές ε, γυναίκες, για εκατομμύρια γυναίκες και παιδιά. Λοιπόν υπάρχουν πάρα πολύ λίγες ευκαιρίες, πάρα πολύ λίγη ασφάλεια, ε, όπως βεβαίως και για πολλούς ε, άντρες. Και βλέπουμε ότι οι αλλαγές στο περιβάλλον μας, στο κλίμα, στη γη που ζούμε έχουν μεγάλες επιπτώσεις στα, στις ανισότητες μεταξύ των φύλων. Από την άλλη, όταν οι γυναίκες έχουν μια ευκαιρία, τότε πραγματικά είναι πολύ σημαντικό ρόλο ώστε να υπάρξει μια καλύτερη και πιο βιώσιμη κοινωνία και πιο δίκαιη. Πολλοί λοιπόν ε, έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ, πολύ, πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, ε, υπάρχουν μεγάλες περίοδοι ξηρασίας, υπάρχουν πολλές πλημμύρες, το επίπεδο της θάλασσας ανεβαίνει. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ μεγάλες απειλές και για το πόσιμο νερό αλλά και για την ε, άρδευση. Και η πολιτική ε, ενέργειας θα πρέπει να ασχοληθεί ακριβώς με, αυτή, με αυτά τα δύο εκατομμύρια ανθρώπων που βασίζονται σε, που ζουν σε τέτοιες ε, δύσκολες συνθήκες. Η ασφάλεια λοιπόν είναι πολύ σημαντική για πολλές κοινότητες και η ασφάλεια είναι όχι μόνο τροφίμων αλλά και νερού, ασφάλεια ε, στέγασης, κατοικίας, ενέργειας. Όλα αυτά σήμερα δυστυχώς διακυβεύονται. Αλλά και η υγεία απειλείται και αυτό συμβαίνει και λόγω των φυσικών καταστροφών αλλά και μέσως, μέσω της επιδείνωσης των συνδικών ζωής. Υπάρχει ελάχιστο πόσιμο νερό, ε, αυξάνονται προφανώς έτσι οι ασθένειες, ελονοσία, κίτρινος πυρετός, όλα αυτά, όλες αυτές οι ασθένειες πλήττουν τους πολίτες ένας ειδικός ε, γιατρός ε, από το Ινστιτούτο, Ερευνητικό Ινστιτούτο της ε, Κένιας, ο Άνδριου Γκιτέκο, είπε ότι τώρα αυτές οι αλλαγές στη θερμοκρασία έχουν οδηγήσει στο να είναι πολύ πιο επιθετικά και τα κουνούπια που μεταφέρουν την ελονοσία. Η IPCC λέει πως οι φτωχές κοινότητες ε, ζούνε σε πολύ συγκεντρωμένες ε, ε, κοινότητες και είναι πάρα πολύ ευάλωτες. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τις συνθήκες αυτές γιατί εξαρτώνται από τα τρόφιμα, από, την, από το νερό, τα οποία όμως επίσης πλήττονται λόγω των κλιματικών αλλαγών. Ε, και θα πρέπει να μπορούν οι κοινότητες αυτές να προσαρμοστούν σε όλε αυτέ τι αλλαγέ και να τι αντιμετωπίσουν. Δυστυχώς όμως ε, για τι φυσικέ καταστροφέ τουλάχιστον δεν έχουν, δεν έχουν κανένα έλεγχο αλλά και για τι κοινωνικέ και για τι οικονομικέ και τι πολιτικέ αλλαγές που συμβαίνουν δεν μπορούν να τι επηρεάσουν. Οι άνθρωποι που ζουν στη φτώχεια πραγματικά είναι πολύ ευαίσθητοι. Ε, πολύ ευάλωτοι οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκε, τα παιδιά, άτομα με ειδικέ ανάγκε, οι μειονότητε, Αυτοί υποφέρουν από τις κλιματικές αλλαγέ. Ένα από τα, από τις, μία από τις μεγαλύτερες ανισότητες στην ε, κοινωνία μας έχει να κάνει με τις κοινωνικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα κορίτσια, έχουν γίνει μικρά βήματα προόδου και στη δική μου τη χώρα, στις κάτω χώρες, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν ε, ακόμα ε, διαφορές ό,τι αφορά τις ευκαιρίες που έχουν τα κορίτσια. Οι κλιματικές αλλαγές δεν είναι ουδέτερες ως προς το φύλλο. Οι γυναίκες είναι αυτές ε, που πλήττονται πολύ περισσότερο από τις κλιματικές αλλαγές. Εδώ βλέπετε κάποιες εικόνες από το Βιετνάμ, ε, γιατί δεν έχουν ε, νερό. Αν δεν έχουν νερό προφανώς πρέπει να αντιμετωπίσουν πολύ, πολλά προβλήματα όταν δεν έχουν τρόφιμα επίσης. Όταν μειώνονται τα τρόφιμα, προφανώ μειώνεται και η ποσότητα που αναλογεί στον καθένα. Και οι γυναίκε επιβαρύνονται και με αυτό. Είναι λοιπόν θύματα από διάφορες, σε διάφορες απειλές, τα κάψιμα μειώνονται, οι γυναίκες επίσης είναι πιο ευαίσθητες σε ό,τι αφορά τις ασθένειες και κυρίως την ελονοσία και ο, η σύνδεση μεταξύ της κοινωνίας και του περιβάλλοντος είναι σημαντική και αυτό φαίνεται και στις κλιματικές αλλαγές τα τρόφιμα και οι καλλιέργειες γίνονται πιο δύσκολες, δεν έχουμε νερό, ε, οι καύσονες γίνονται όλο και πιο έντονοι, οι φυσικές καταστροφές είναι και πιο πολλές, βλέπουμε και στο Μπαγκλαντές τι γίνεται, υπάρχουν και μελέτες από το LSE όπου λέει ότι υπάρχουν, έχουν υπάρξει 140 φυσικές καταστροφές πρόσφατα και οι γυναίκες έχουν όλο και λιγότερες πιθανότητες να επιβιώσουν. Οι μεγαλύτερες όσο μεγαλύτερη είναι η καταστροφή, τόσο μεγαλύτερη συνέπειε έχει και τόσο πιο πολύ πλήττει αυτή την ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Και πλήττει βεβαίω κυρίω τι γυναίκε. Βεβαίω υπάρχουν περιπτώσει όπου πλήττονται περισσότερο οι άντρε, αλλά αυτό είναι πιο σπάνιο το Μπαγκλαντές, το Άτσε, η Ινδονησία, είδαμε ότι από 55% 70% γυναίκες ήταν τα θύματα από το τσουνάμι ήδη από το 2004. Οι γυναίκες που είναι φτωχές και χάνουν ό,τι υπάρχοντα έχουν, καταλήγουν να ζουν με, με, με μηδενικούς πόρους. Ο τυφώνας Κατρίνα, στη Λουιζιάννα και στο Μισισίπι, στις Ηνωμένε Πολιτείες έπληξε πάρα πολύ τις ε, γυναίκες ε, τις Αφροαμερικανίδες. Αυτές είναι η πιο ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα και αυτό δείχνει και πόσο σημαντική είναι ε, πόσο σημαντικές είναι αυτές οι συνέπειες. Γιατί δεν μιλούμε μόνο για το φύλλο, αλλά μιλούμε και για την εθνοτική προέλευση και για την ηλικία και για το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο του καθενό. και έτσι φαίνεται πόσο ευαίσθητες ε, ευάλωτες είναι οι γυναίκες. Στο Βιετνάμ οι γυναίκες είναι τα θύματα. Στις περιπτώσεις που μελέτησα εγώ, οι γυναίκες με κάποιο τρόπο οργανώθηκαν, ήταν, έγιναν ακτιβίστριες, προσπάθησαν ε, να αντιμετωπίσουν, να λύσουν τα προβλήματα του περιβάλλοντος, να δημιουργήσουν και πάλι τις κοινότητές τους. Η Σαχίνα Ντεγκούν ζει σε ένα χωριό στο Μπαγκλαντές όπου υπάρχουν συνεχείς πλημμύρες. Δεν αισθάνεται όμως, δεν αισθάνεται θύμα, λέει ότι ε, δεν ε, γεννηθήκαμε για να υποφέρουμε, λέει γεννηθήκαμε για να παλεύουμε. Και η η ε, Σαχένα ε, όταν δεν είχε ε, τελειώσει ακόμα το σχολείο όταν αποφάσισε να κάνει, ένα, να κάνει μαθήματα για την αντιμετώπιση των κρίσεων και τώρα είναι πρόεδρος της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των κρίσεων και εξήγησε στις γυναίκες πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν μια τέτοια καταστροφή. Ας πούμε το ξύλο το, διατηρούμε, το διατηρούν πλέον οι γυναίκες σε υψηλότερα σημεία που δεν μπορεί να τα φτάσει το νερό. Τα τρόφιμα επίσης. Οι γυναίκες λοιπόν πλέον είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια καταστροφή. Επίσης, μιλήσαμε για τους ε, πρόσφυγες λόγω των κλιματικών αλλαγών και για τη μετανάστευση. Το θέμα αυτό είναι πολύ περίπλοκο και μάλιστα μια... Ε, ε, εφημερίδα ε, στις, στις ε, κάτω χώρες είπε ότι θα υπάρξουν 50 εκατομμύρια πρόσφυγες μέχρι το 2015. Επίσης το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας είπε ότι όταν κάποιος πρέπει να ζήσει κάτω από άσχημες συνθήκες, προφανώς φεύγει από τη χώρα του, μεταναστεύει για να βρει μια καλύτερη ζωή και συνήθως είναι οι γυναίκες αυτές που φεύγουν. Υπάρχουν ε, ε, πλημμύρες, υπάρχουν φυσικές καταστροφές, ε, υπάρχουν ανεμοστρόβιλοι που συνέχεια βλέπουμε άρθρα για όλα αυτά στις στις εφημερίδες, βλέπουμε άρθρα για, τις, για την ξηρασία και η ξηρασία θα είναι ένα από τα βασικά προβλήματα για τις γυναίκες στο μέλλον. Εγώ κατανοώ ότι πολλές γυναίκες μετά από φυσικές καταστροφές θέλουν να αντιδράσουν, θέλουν να δημιουργήσουν κοινωνικά δίκτυα, θέλουν να κινητοποιηθούν, το έχω πει. Οι άντρες συνήθως φεύγουν, ψάχνουν έναν άλλο, ένα άλλο σπίτι, μια άλλη δουλειά και διαπιστώνει κανείς ότι οι γυναίκες μένουν πίσω και προσπαθούν να προστατεύσουν την, την οικογένειά τους. Αυτό είναι ένα επιπλέον βάρος λοιπόν για τις γυναίκες. Όταν φεύγουν, όταν μεταναστεύουν οι γυναίκες, τότε αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερους ε, κινδύνους. Η International Plan ε, από το Ηνωμένο Βασίλειο είπε, ε, παρατήρησε πολλές ε, τέτοιες περιπτώσεις στον Παγκλαντές και την Αιθιοπία για τις ε, ε, επιδεινωμένες ε, συνθήκες επιβίωσης και που οδήγησαν τις γυναίκες στο να παντρεύονται νωρίς για να έχουν κάποιο στήριγμα ή να οδηγούνται στην πορνεία. Υπάρχουν λοιπόν πάρα, πολλές, πάρα πολλοί κίνδυνοι. Οι συνθήκες λοιπόν είναι πολύ διαφορετικές. Το πώς πλήττουν οι κλιματικές συνθήκες της, τους άντρες και τις γυναίκες είναι πολύ διαφορετικό. Λοιπόν, προσπάθησα να σας παρουσιάσω τις ε, κοινωνικές συνέπειες των ε, ε, κλιματικών αλλαγών και κυρίως το πώς αυτές επηρεάζουν τις, τα δύο φύλλα. Είναι σημαντικό οι επιστήμονες και οι πολιτικοί να αναγνωρίσουν ότι οι κλιματικές αλλαγές δεν είναι μόνο τεχνικό και πολιτικό θέμα σε, που πλήττει όλους σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα στην πολιτική, στα προγράμματα, στα ε, projects που υπάρχουν, θα πρέπει αυτά τα, αυτές οι πιο ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες να τύχουν της απαραίτητης προστασίας και σε ό,τι αφορά την, ε, την αντιμετώπιση αυτή καθ' αυτή των κλιματικών αλλαγών, αλλά και σε ό,τι αφορά την απώλεια της ασφάλειας που νιώθουν πια. πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε και για τις γυναίκες και για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους και κυρίως πρέπει να προστατεύσουμε τους φτωχούς και τους μετανάστες σε όταν εκπονούμε νέες πολιτικές. Αυτή λοιπόν είναι η... Αυτή είναι η κοπέλα που σας έλεγα, η Χαγκάρη Ματάη από την Ινδία με τον αδερφό της και για αυτή είναι η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε ο ε, Έχουμε κάποια τεχνικά προβληματάκια. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Πολύ ενδιαφέροντα. Αναφερθήκατε, ε, αγαπητή Ρέν Ντάγκελμαν, σε πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά πράγματα. Και βλέπουμε βεβαίως ότι οι γυναίκες δεν είναι μόνο θύματα, είναι και μέρη της λύσης και συμφωνώ απολύτως με την τοποθέτησή σας. Συνεχίζουμε λοιπόν και θα δώσουμε αμέσως το λόγο στην Ιωάννα Μπόρτσα, η οποία είναι εμπειρογνώμων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων Ε, και θα μας κάνει τη δική της εισήγηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση. Πρέπει να σας πω ότι από τεχνικής απόψεως είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό ε, Ιστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, που είναι ένα σχετικά νέο Ινστιτούτο, παρουσιάζει εδώ ενώπιόν σας την εργασία του. Και χαίρομαι που είμαι εγώ αυτή που θα κάνει την πρώτη παρουσίαση. Τίτλος της παρουσίασής μου, στην οποία θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομη, μια και πολλά σημεία τα οποία θέλω να θίξω θίγησαν ήδη, είναι φόκους για την Ευρώπη του 2012 ξεκινώντας από τον ε, Ιανουάριο του 12 με την Δανέζικη Προεδρία δηλαδή ε, στα πλαίσια της Προεδρίας ε, εστίαση θα δοθεί εις τη θέση των γυναικών και την ισότητα των φύλων απέναντι στην κλιματική αλλαγή και εμείς προετοιμάζουμε το έγγραφο της Προεδρίας υλοποιώντας βεβαίως και το σχέδιο της Βελγικής Προεδρίας την πλατφόρμα σκέψης κλπ. Τα κύρια σημεία τα οποία θα παρουσιάσω σήμερα απορρέουν ακριβώς από αυτήν την ε, μελέτη και την προετοιμασία που κάναμε ε, για να εκπονήσουμε την μελέτη αυτή. τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου θα είναι όλα έτοιμα. Μετά θα ξεκινήσει και η ε, διοικητική ας πούμε, διαδικασία και ελπίζουμε ότι Φεβρουάριο, αρχές Μαρτίου θα δημοσιευθεί και θα είναι διαθέσιμη για όλους. One of the aims of this... Ένας από τους στόχους λοιπόν αυτής της ε, έκφρασης ε, και αφορά ακριβώς τις γυναίκες απέναντι στην κλιματική αλλαγή, αλλά ε, ξεκινούμε επικεντρωνόμενοι στην ε, Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. αλλά βεβαίως ε, προσεγγίζουμε το θέμα με την ε, προοπτική της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, βλέποντας όμως τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν το ζήτημα ε, και πώς ε, αντιμετωπίζουν στην Ευρώπη την κατάσταση της κλιματικής αλλαγής. Okay, the main, the main topics that I would, will address. Τα κυριότερα στοιχεία τα οποία ε, θα αντιμετωπίσουμε εδώ είναι αυτά που βλέπετε γραμμένα στη διαφάνεια, κυρίως δηλαδή πώς πώς ε, μπορούμε να δούμε από ε, σκοπιά ισότητας φύλων, από πλευρά ε, κινητικότητας, πώς οι άνδρες και οι γυναίκες από διαφορετικές οπτικές γωνίες μπορούν να συμβάλλουν ή συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Δεν θέλουμε να καταμερίσουμε ευθύνε ή να κατηγορήσουμε τους μένιν τους δε, προσπαθούμε να υπογραμμίσουμε αυτά τα θέματα και να οδηγήσουμε κατά κάποιο τρόπο με τα συμπεράσματά μας σε τις πολιτικές οι οποίες θα αναπτυχθούν. Επίσης προσπαθούμε να βρούμε ποιε είναι οι διαφορετικές ικανότητε που έχουν οι άντρε και οι γυναίκες και ε, ε, με πιο διαφορετικό τρόπο ανταποκρίνονται ε, στις διάφορες απειλές που προκύπτουν από τις αλλαγές του κλίματος. Να δούμε λοιπόν πώς βλέπει είναι οι άνδρες και οι γυναίκες στην κλιματική αλλαγή ε, και με ποιο τρόπο μπορούμε να ε, ε, εμπνευστούμε κατά κάποιο τρόπο από τα στοιχεία αυτά στην υλοποίηση πολιτικών. Όσον αφορά την έρευνα για την κλιματική αλλαγή, ε, η θέση των γυναικών δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολύ ε, ψαχτεί κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένα δευτερεύον, να το πούμε, αλλά παρόλα αυτά ε, εμεί θεωρούμε ότι η θέση των φίλων απέναντι στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών δεν πρέπει να περιθωριοποιείται. Δεν υπάρχει επίσης μεγάλη πολύ αναπτυγμένη έρευνα ε, όσον αφορά τα θέματα αυτά γιατί ε, οι μελετητές ε, δεν έχουν σκύψει με μεγάλο ενδιαφέρον φαίνεται πάνω σε αυτό το θέμα γιατί δεν είναι ελλειπής και η πόρη η χρηματοδότηση των ερευνών αυτών, των, των μελετών αυτών. Εμείς προσπαθούμε λοιπόν είπαμε, να βάλουμε τη διάσταση των, του φύλου στις ε, ε του κλίματος και λέμε ότι ε, θα πρέπει να λάβουμε, να αντιμετωπίσουμε μάλλον την κλιματική αλλαγή ε, σαν θέμα κοινωνικής ευθύνης, ανθρώπινης ευγένεια, σαν οικουμενική υποχρέωση. Θα ήθελα ε, εντάχει να πω κάτι γιατί αναφέρθηκε ήδη προηγουμένως ε, λόγω των διαφορετικών ρόλων που έχουν στην κοινωνία οι άνδρες και οι γυναίκες ε, ε, λόγω της διαφορετικής πρόσβασης ε, που ε, έχουν στο κοινωνικό στάτους, στην εκπαίδευση, στα, στους πόρους κτλ. Με τον ίδιο τρόπο και αντίστοιχα η επιπτώση από την αλλαγή μπορεί να διαφέρει είχαμε μία έρευνα στην περιοχή της Αρκτικής και εκεί κατεδείχθη ότι ότι οι γυναίκες, ότι γενικά οι ανθρώπινοι πληθυσμοί που είναι εγκαταστημένοι εκεί αντιμετωπίζουν διαφορετικά τις κλιματικές αλλαγές. Οι γυναίκες φαίνεται ότι ε, προσαρμόζονται καλύτερα στην ε, νέα κατάσταση αλλά ε, καλύτερα από τους άντρες. Εδώ δεν επαναλαμβάνω ότι δεν, δεν γίνεται καταμερισμός ευθυνών ή θέλουμε, δεν θέλουμε να πούμε ότι ε, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Απλώς βλέπουμε ότι ε, ε, αντιμετωπίζουν διαφορετικά τις πλημμύρες, τις ξηρασίες, οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή τους. Όσον αφορά τώρα τις εκπομπές το, του φαινομένου του θερμοκηπίου, λόγω και του κοινωνικού τους ε, στάτους οι άνδρες ε, χρησιμοποιούν περισσότερο τεχνολογίες, ε, κυκλοφορούν περισσότερο, επομένως παράγουν κατά κάποιο τρόπο περισσότερους ρήπους, περισσότερα αέρια τα οποία συμβάλλουν στο φαινόμενο της, του θερμοκηπίου, ενώ οι γυναίκες μένουν περισσότερο στο σπίτι, μεγαλώνουν τα παιδιά τους κτλ. Ε, επίσης όσον αφορά την διατροφή ε, είναι γεγονός ότι οι άνδρες και λόγω Comparative in λόγω των σωματικών τους αναγκών καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες τροφής. Uh, sex, gender, uh, και συμβάλλουν επομένως περισσότερο σε, αυτήν την, ε, σε αυτό το σύστημα διατροφικής αλυσίδας. Ε, η πρόσβαση στους πόρους, η πρόσβαση ε, στα επαγγέλματα επίσης διαφέρει από τους άνδρες και γυναίκες και επομένως έχουν διαφορετική προσέγγιση άνδρες στις γυναίκες. Διαφορετική προσέγγιση επίσης υπάρχει ε, και όσον αφορά την, τον μετριασμό της επίπτωσης των κλιματικών αλλαγών. Τα αγόρια και τα κορίτσια δεν έχουν απαραίτητα ε, και πάντοτε και σε όλα τα επίπεδα ίδια ε, δυνατότητα πρόσβασης ε, στην εκπαίδευση ούτε άλλωστε ίδιες αμοιβέ. Αυτή η κατάσταση θα έχει αντίκτυπο στην καθημερινή του ζωή και στην καθημερινή τους ε, ε, ενασχόληση. Ε, ας πούμε δεν θα επιλέξουν απαραίτητα ε, μια πιο πράσινη τεχνολογία ή έναν ε, πάροχο ενέργειας που σέβεται περισσότερο το περιβάλλον γιατί δεν έχουν τις γνώσεις ενδεχομένως να το κάνουν και επομένως λόγω έλλειψης και γνώσεων μπορεί να μην είναι τόσο τόσο ευαίσθητες όσον αφορά ε, την ε, χρήση πράσινων, πράσινης ενέργειας. αντιλήψεις και στάσεις ε, απέναντι στην, στον μετριασμό των αντικτύπων της κλιματικής αλλαγής. Εδώ ενδεχομένως είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Υπάρχει το Ευρωβαρόμετρο που πρόσφατα ε, εξεπώνησε μελέτη αλλά και γενικώ υπάρχουν ε, αποδεικτικά στοιχεία ε, βάσει του οποίου τεκμηριώνονται οι διαφορές ανάμεσα στην αντίληψη που έχουν οι άνδρες και οι γυναίκες και τη στάση που έχουν απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Ε, καταδεικνύεται σαφώς η σημασία ε, του ε, θέματος αυτού και σε ορισμένα κράτη-μέλη ήδη έχουν προχωρήσει περισσότερο οι μελέτες και γίνεται μια προσπάθεια να μελετηθούν από κοντά οι διαφορές. Οι γυναίκες φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την κλιματική αλλαγή ως μεγαλύτερη απειλή Επίσης ε, είναι κατά της ε, πυρηνικής ενέργειας ε, ή κάποιων επιθετικών μορφών ενέργειας γιατί πιστεύουν ότι θα επιβαρύνουν περισσότερο τις κλιματικές αλλαγές. Το γεγονός ότι φροντίζουν τα παιδιά επίσης τις κάνει πιο ευαίσθητες απέναντι σε τέτοια θέματα ε, και σε τεχνικές λύσεις οι οποίες ε, θα βελτιώσουν ε, την κατάσταση του πλανήτη. Αλλά και εδώ βέβαια παρεμβαίνουν παράγοντες που ανέφερα προηγουμένως η έλλειψη κατάρτισης γνώσεων κτλ τα διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από τις διάφορες κυβερνήσεις όσο αμφισβητήσιμα και κι αν είναι τα αριθμητικά στοιχεία, ε, γιατί βεβαίω αυτά μπορεί κανεί να τα συζητήσει, αλλά παρόλα αυτά εμεί προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο ε, οι διάφορε στρατηγικέ αντιμετώπιση και πολιτικές αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και προβλημάτων μπορούν να έχουν αντίκτυπο διαφορετικό στι άντρε και στι γυναίκε. υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία οι γυναίκες θεωρούν ε, ε, ότι τις απασχολούν περισσότερο. Ας πούμε, οι δημοσιονομικές ε, ρυθμίσεις, φόροι, τρόπος φορολόγησης της ενέργειας κτλ. Ε, ε, εδώ προσπαθώ να αναφερθώ την ανάγκη να υπάρξει το ερώτημα ε, της ισότητας ε, απέναντι στις κλιματικές αλλαγές. Είπαμε ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές προοπτικές, ε, όχι μεταξύ των ανδρών και των γυναικών μόνο, αλλά και μεταξύ των ιδίων των γυναικών. Στα ίδια τα κράτη-μέλη ή μεταξύ διαφόρων κρατών μελών, μεταξύ διαφόρων περιοχών των ιδίων κρατών μελών υπάρχουν αλλαγές οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν αντιμετωπίζουμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Δεύτερη παύλα για το γιατί θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισότητα των φίλων για μα γιατί είναι θέμα δικαιοσύνης, είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Και η λήψη αποφάσεων που μας επηρεάζει όλους θα πρέπει να λάβει υπόψη ε, διαφορετικές οπτικές γωνίες, διαφορετικούς τρόπους έκφρασης, ε, ιδιαιτερότητες και βεβαίως είναι και θέμα, αξι... Ε, και, θέμα αποτελεσματικότητας. Ε, το σημαντικό είναι να βρούμε λύσεις ε, για τα προβλήματα τα οποία όλοι αντιμετωπίζουμε, λαμβάνοντας όμως υπόψη και τις ιδιαιτερότητες ε, ορισμένων ομάδων. Όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποιος παίρνει τις αποφάσεις, με ποιο τρόπο, με, ποια, με ποιο οικονομικό υπόβαθρο κτλ. κτλ επίσης τους ε, διάφορους τρόπους ε, με τους οποίους βλέπουμε την κλιματική αλλαγή, δηλαδή πώς λαμβάνουμε, πώς, ε, πώς, παίρνουμε, πώς επιλέγουμε τους τελικούς τις τελικές στρατηγικές και πολιτικές, πώς επιλέγουμε τους στόχους κτλ. Θα επανέλθω στο σημείο από το οποίο ξεκίνησα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ισότητας των φύλων. Θέλω να πω ότι θα πρέπει σοβαρά να λάβει υπόψη την ισότητα των φύλων για όλους τους λόγους που εξήγησα πριν. Eh, Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση. Κυρία Μπόρζα. Και είναι να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Συνισότητα των Φύλων, στο οποίο εργάζεστε. Είναι πολύ χρήσιμο για εμάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι μας διευκολύνει, μας προσφέρει στατιστικά στοιχεία, δείκτες, κάνει μετρήσεις και έρευνες και μας επιτρέπει να λαμβάνουμε καλύτερες αποφάσεις. Θα δώσω το λόγο στη Σκιώδη συγγήτρια, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Νικόλ Κιλ Νίλσεν για ένα σχόλιο ή μια ερώτηση, δεν ξέρω. Ναι, θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα στην κυρία Επίτροπο και να μας πει αν πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Το γεγονός ότι η λέξη «φίλο» η λέξη γυναίκες δεν εμφανίζεται ποτέ. Είναι λέξεις που δεν εμφανίζονται ποτέ στα, ευρωπαϊκό, στα ευρωπαϊκά κείμενα για την, ε, για την κλιματική αλλαγή, όπως είναι η στρατηγική για την Ευρώπη το 2020, μεταξύ άλλων. Ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα και να εμφανιστούν οι όροι αυτοί, φίλο ή οι γυναίκες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τη διάσταση του φύλου, θα αρχίσει να συλλέγει δεδομένα φύλο. θα υλοποιήσει φιλόδοξα προγράμματα ούτως ώστε να ε, διάφοροι τομείς να προσελκύσουν ε, περισσότερες γυναίκες. Το είδαμε με την ε, πρωτοβουλία που αναλήφθηκε πριν από κάποια χρόνια ώστε να ενθαρρύνονται τα κορίτσια να κατευθύνονται στις σπουδές και στα εργασιακά ε, προς ε, τον τομέα της μελλοντική πράσινης οικονομίας. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος θέλει να κάνετε σχόλιο. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ. Yes, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι ο, ο... ότι όντως η λέξη φύλλο δεν αναφέρεται στο 21ο πρόγραμμα και το καθεξής, το roadmap δηλαδή. Δεν θα σας πω ότι ναι, την επόμενη φορά που θα σας δω θα αναφέρεται και θα έχει συμπεριληφθεί. Πολλά πράγματα πρέπει να συμπεριληφθούν στο roadmap και δεν θέλουμε να ε, φύγει το σημείο εστίασης ε, και να ε, γίνει πιο έκεντρο. Μας ενδιέφερε περισσότερο στο roadmap, στον οδικό χάρτη, η μετατροπή των πηγών ενέργειας σε πιο πράσινες πηγές ενέργειας, ε, η αλλαγή της πολιτικής και ε, όλων αυτών που πρέπει να κάνουμε σε επίπεδο κτηρίων, σε επίπεδο γεωργίας και το καθεξής. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που ακούστηκε από την προηγούμενη ομιλήτρια για τα θέματα φορολόγησης. Εγώ είμαι υπέρ μιας πιο πράσινης φορολόγησης. Ωστόσο, όταν ε, επιβάλλουμε πράσινη φορολόγηση, θα πρέπει να δούμε και ποιο θα είναι το αντιστάθμισμα και σε επίπεδο κτηρίων και άλλων. Βέβαια πολλά είναι τα θέματα που επισέρχονται εκεί. Και συμφωνώ απολύτως με την ε, κυρία ε, Κιλ Νίλσεν για τα δεδομένα και τα αριθμητικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα δύο φύλλα. Όταν ε, μπορούμε να συλλέξουμε όσο τα περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για όλα τα θέματα, πληροφορίες δηλαδή για το πώς εκπροσωπούνται τα φύλλα, τα δύο φύλλα, αυτό μας βοηθά γιατί λαμβάνουμε πιο ενημερωμένες αποφάσεις και ξέρουμε πολύ καλύτερα ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από τις αποφάσεις μας. Έτσι είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε αποφάσεις με τα λόγου γνώσης. Επομένως όντως πρέπει να έχουμε περισσότερα στοιχεία για, το, για την ισότητα των φύλων. Ευχαριστώ. Θέλετε να προσθέσετε και κάτι άλλο. Εάν όχι, πολύ ωραία. Θα συνεχίσουμε τώρα. Έχουμε λοιπόν σύντομα σχόλια από πλευράς ε, μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ξεκινήσουμε με τη σκιώδη συγγήτρια ή την κυρία Στρέλα πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομη. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τις ομιλήτριες για τα παραδείγματα για τις έρευνες, τις μελέτες, τα γεγονότα, τα ποσοστά, τα αριθμητικά στοιχεία που παρουσίασαν. Εγώ ήμουν εισηγήτρια μιας έκθεσης για την κλιματική αλλαγή και έχω συμμετάσχει σε πολλές ε, διασκέψεις και σε πολλά συνέδρια για την ε, κλιματική αλλαγή εν γέννη. Και στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών ασχολούμαι με τα θέματα των διακρίσεων όπου τα θύματα είναι γυναίκες. Και σε αυτή την έκθεση θα προσπαθήσω να συνοψίσω αυτές τις δύο βασικές αγωνίες μου, αν θέλετε, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σαφές ότι οι γυναίκες πλήττονται ε, περισσότερο από τις δύσκολες καταστάσεις. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας, διότι πρόκειται για μια κοινωνική ομάδα η οποία υφίσταται ε, διακρίσεις. Για παράδειγμα η κρίση που έχουμε σήμερα δεν είναι οι γυναίκες ο βασικός υπέτειος ε, της χρηματοοικονομικής κρίσης που μας οδήγησε στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Ωστόσο, είναι οι γυναίκες τα βασικά θύματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το ίδιο συμβαίνει και με τους κατακλυσμούς, τις φυσικές καταστροφές, καταστροφές το ίδιο συμβαίνει και με τη φτώχεια και ούτω καθεξής. Οι γυναίκε, λοιπόν Ε, είναι μια κοινωνική ομάδα που πάσχει περισσότερο από αναλφαβητισμό, έχει λιγότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση, στην εκπαίδευση, στην παιδεία. Δεν γνωρίζει πολύ συχνά τα δικαιώματά της, έχει λιγότερη οικονομική ισχύ, απολαμβάνει λιγότερο κοινωνικό κύρος, η κοινωνική αυτή ομάδα των γυναικών. Καταλαμβάνουν θέσεις απασχόλησης με μικρότερη αμοιβή, οι θέσεις απασχόλησης που δεν ε, χαίρουν τόσο μεγάλου κύρους. Ε, Πολύ συχνά οι γυναίκες μπορεί να είναι θύματα ε, προκαταλήψεων ε, θρησκευτικών, πολιτισμικών ή άλλων. Και είναι οι γυναίκες αυτές που ενδιαφέρονται κυρίως για, την, για το καλό επίπεδο ζωής και τα προβλήματα των παιδιών τους και των οικογενειών τους γενικότερα. Είναι οι τελευταίες που τρώνε φυσικά όταν υπάρχει έλλειψη τροφίμων. Επιπλέον, οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια. Εάν υπάρχει περίπτωση να ε, ξεσπάσει κάποια στιγμή στο μέλλον τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, τότε σίγουρα αυτός θα ήταν ο πόλεμος για το νερό και για τα τρόφιμα. Και αν γινόταν κάτι τέτοιο, είναι βέβαιο ότι πάλι τα μεγαλύτερα και τα περισσότερα θύματα θα ήταν γυναίκες. Και έχουμε σήμερα βεβαίως και τους πρόσφυγες για κλιματικούς λόγους, για λόγους κλιματικής αλλαγής. Είναι μια νέα κατηγορία προσφύγων και η πλειονότητα εξαφών είναι γυναίκες. Παρόλα αυτά, οι γυναίκες δεν συμμετέχουν επαρκώς στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Δεν συμμετέχουν στις αποφάσεις για το μετριασμό και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή ε, στην κλιματική αλλαγή. Θα έλεγα μάλιστα ότι έχουν μεγάλη ευθύνη στη διαχείριση φυσικών πόρων οι οποίοι είναι ελάχιστοι και λόγω αυτής της συμμετοχής τους ε, σε αυτή τη δραστηριότητα γνωρίζουν πολλά περισσότερα και είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένες. Ε, όταν γίνεται λόγος για την περιβαλλοντική αηφορία. Εξού και έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν στην πρόληψη των φυσικών ε, καταστροφών, κάτι το οποίο είναι θεμελιώδες για την ε, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Θα ήθελα επίσης να συμπληρώσω το εξής. Αναμφίβολα, η δημοκρατία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η επίτευξη ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών θα συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος ε, και στο καλύτερο μέλλον για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, και εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Γιανακουδάκη. Παρακαλώ. Ζω ότι οι γυναίκες είναι ισχυρές είναι ικανές, μπορούν να προσφέρουν έργο. Δεν έχουν επίσημη, αν θέλετε, εκπαίδευση, αλλά μπορούν να σταθούν επάξια απέναντι σε έναν άντρα. Νομίζω ότι είμαστε ίσες έναντι των ανδρών και δεν θα δεχθώ ε, αυτή την εικόνα της κακομήρας γυναικούλας η οποία είναι στριμωγμένη στη γωνία. Αυτό γενικά σαν γενική παρατήρηση. Από εκεί και πέρα. Στο θέμα μας τώρα, οι κλιματικές αλλαγές. Στην αρχή δυσκολεύτηκα να καταλάβω γιατί είναι θέμα που ε, αφορά ιδιαίτερα τις γυναίκες και γιατί θα πρέπει να το εξετάζουμε από την οπτική γωνία των γυναικών. Δεν μ' αρέσει να καταλήγουμε σε στερεότυπες εικόνες των ε, γυναικών. Είπε κάποια ομιλήτρια που ότι ελέγχουν καλύτερα τον οικοκυριό τους ή τις εκπομπές αν θέλετε ε, του οικοκυριού τους. Ναι, μπορεί αυτό να ισχύει ότι έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν πιο οικολογικά προϊόντα ή λιγότερο. Μπορεί κανείς να πει ε, ότι οι γυναίκες είναι αυτές που βασικά εκπαιδεύουν την επόμενη γενιά, επομένως είναι σε θέση να έχουν μια πιο πράσινη προσέγγιση και να τη μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά τους. Αυτό το δέχομαι και ισχύει. Ωστόσο, Είπε, κάποιος, είπε κάποια από τις ομιλήτριες ότι δεν είναι τόσο ευαίσθητες όταν κάνουν επιλογές. Για παράδειγμα, όταν επιλέγουν το αυτοκίνητο. Εγώ νομίζω ότι έχουν διανύσει μεγάλη απόσταση οι γυναίκες, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη λοιπόν οι γυναίκες διαλέγουν οι ίδιες το αυτοκίνητό τους και διαλέγουν ένα πιο πράσινο αυτοκίνητο όταν έχουν την οικονομική αυτή δυνατότητα. Διότι τα πράσινα αυτοκίνητα είναι κάπως πιο ακριβά από τα υπόλοιπα μέχρι αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα λοιπόν ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις και σε πάρα πολλές καταστάσεις οι γυναίκες όντως είναι υπεύθυνε γιατί εν γέννη αυτές ε, κρατούν τα ενία του νοικοκυριού όχι γιατί δεν δουλεύουν αλλά γιατί πολύ συχνά κάνουν και τα δύο και όντως μπορούν να εκπαιδεύσουν και εκπαιδεύουν την επόμενη γενιά, όντως είναι πιο ευαίσθητες διότι αντιλαμβάνονται την εμπλοκή των άλλων ομάδων, των κοινωνικών και πρέπει να τις συμπεριλάβουμε τις άλλες κοινωνικές ομάδες όταν γίνεται λόγος για ε, κλιματική αλλαγή για να μην έχουμε πολλαπλές ανισότητες. Από εκεί και πέρα η πρώτη ομιλήτρια μίλησε για το πόσο οι γυναίκες πλήττονται στις χώρες του τρίτου κόσμου και είναι κάτι το οποίο βλέπω όντως. Οι γυναίκες στις περιοχές αυτές έχουν την τάση να είναι κατά τη φτωχότερες από τους ε, άνδρες και χρειάζονται περισσότερο η στήριξη ε, στη γεωργία, σε διάφορες δραστηριότητες για να αυξήσουν το εισόδημά τους. Εν τούτης, το ερώτημα η κλιματική αλλαγή πλήττει τις γυναίκες μόνο ή κατά κύριο λόγο. Εγώ θα έλεγα ότι πλήττει τους πάντες και πρέπει να υιοθετήσουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση. Ε, δεν ξέρω αν είναι θέμα που έχει να κάνει με τη διάσταση του φύλου. Η διάσταση του φύλου είναι μία από τις συναισθώσεις. Είναι κοινωνική και ανθρώπινη ευθύνη. Κάποια από τις ομιλήτριες το είπε αυτό και συμφωνώ απολύτως. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πάμε. Καλό είναι που συζητούμε δηλαδή ε, το θέμα αυτό υπό την ε, οπτική γωνία ε, της ισότητας των δύο φύλων, αλλά να γνωρίζουμε ότι είναι κάτι το πολύ πιο ευρύ. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος και εγώ ευχαριστώ. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, Ιρένε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια και τις παρεμβάσεις σας δείχνει πόσο θέλετε να εμπλακείτε στο ζήτημα αυτό η κάθε μία από τις σκοπιά της και αυτό είναι πολύ θετικό. Να απαντήσω σε αυτό που είπε η προηγούμενη μιλήτρια και να αποδείξω γιατί είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με τη διάσταση των φύλων. Οι περιβαλλοντικές αλλαγές και οι κλιματικές αλλαγές αυξάνουν και οξύνουν τις κοινωνικές ανισότητες και τις κοινωνικές διαφορές και η πιο σαφή σαφής κοινωνική ανισότητα στον κόσμο είναι η ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Επομένως, εάν δεν αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές με τρόπο κάτω τον οποίο να απαλύνουμε και να εξαλείψουμε τις κοινωνικές αυτές ανισότητες, διατρέχουμε τον κίνδυνο να τις οξύνουμε. Είναι δηλαδή ένα κίνητρο αυτό. Είναι απαραίτητο να δούμε όλες αυτές τις διαφορές. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άλλου είδους ε, κοινωνικές διαφορές και ε, τα έχουμε όλα αυτά ε, ε, συζητήσει. Μιλούμε για το πόσο υπάρχει αλληλοσύνδεση, αλληλοσύνδεση μεταξύ φτώχειας και ανισότητας, αλληλοσύνδεση μεταξύ φτώχειας και AIDS π.χ. Ποια είναι η διαφορά να μεγαλώνει ένα κορίτσι σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας και ποια είναι η διαφορά να μεγαλώνει ένα αγόρι σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Σίγουρα είναι θέματα όλα αυτά που πρέπει να εξετάσουμε και το λέω καταρχάς για να απαντήσω στην προηγούμενη ομιλήτρια και όντω οι γυναίκες πλήττονται. Ωστόσο δεν είναι μόνο ε, πληγήσει, είναι και μεγάλοι ε, παράγοντες δράσης ε, σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ η κυρία Μπόρζα. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτά τα σχόλια, για τις διαφορετικές προοπτικές, τις δικές σας που μας παρουσιάσατε. Θα ήθελα να σχολιάσω την παραδοχή η οποία θέλει τις γυναίκες να είναι θύματα. Όντως πολύ συχνά όταν γίνεται λόγος για κλιματική αλλαγή λέμε ότι οι γυναίκες είναι ε, θύματα της κλιματικής αλλαγής και έχουν τεθεί σε μια πολύ ευπαθή θέση και το καθεξής. Ωστόσο, γίνεται προσπάθεια να δείξουμε πόσο εμπλέκονται και σε άλλα επίπεδα επίσης που έχουν να κάνουν με το ευρύτερο αυτό θέμα. Έχουν λύσει στα χέρια, στα χέρια τους. Νομίζω ότι αντισταθμίζεται αυτή η αρνητική παραδοχή του να θυματοποιούμε τις γυναίκες όταν τονίζουμε ε, και την εμπλοκή τους ε, σε άλλα πράγματα, στη γνώση που έχουν για παράδειγμα για ε, το βιώσιμο τρόπο διαβίωσης. Αυτό το οποίο λείπει είναι η συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πώς έχουν περισσότερη πρόσβαση στη διαδικασία αυτή. Αυτά θα πρέπει να τα προσέξουμε και να τα τονίσουμε. Από εκεί και πέρα ως προς το παράδειγμα του αν η γυναίκα επιλέγει το αυτοκίνητο που θα έχει ε, ένα νοικοκυριό, μια οικογένεια ή αν είναι πιο υπεύθυνη για την καθημερινότητα των μελών της οικογένειας. Τα προβάλαμε όλα αυτά ως επιχείρημα για να δείξουμε ότι λόγω αυτών των ανησυχιών και λόγω όλων αυτών αυτών των πραγμάτων που έχουν οι γυναίκες στο κεφάλι τους καθημερινά, πολύ συχνά δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να αγοράσουν π.χ. ένα πιο οικολογικό αυτοκίνητο ή να κάνουν τέτοιου είδους επιλογές. Οφείλουν λοιπόν οι πολιτικές να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις δυσκολίες των γυναικών, να τις ενημερώνουμε περισσότερο και να τους δίνουμε περισσότερες δυνατότητες, παρά να λέμε ότι δεν το ξέρουν το θέμα ή ε, δεν κάνουν τις σωστές επιλογές. Δηλαδή να είμαστε επικοδομητικοί. Το επιχείρημα το παρουσιάσαμε για να ε, υιοθετήσουμε πιο οικοδομητική στάση. Η Επίτροπος θα πρέπει να φύγει να της δώσω το λόγο για τα τελευταία σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι σε αυτή τη συζήτηση πρέπει να διαφοροποιήσουμε την κλιματική αλλαγή και τις γυναίκες στην Ευρώπη και το ίδιο πράγμα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος οξύνει τις υφιστάμενες ανισότητες. Σε ορισμένες χώρες, είτε είναι η Σομαλία, είτε το Μπαγκλαντές, είτε το Βιετνάμ, είτε αλλού, είναι αναφίβολο το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει διαφορετικά τα δύο φύλλα λόγω της διαφορετικής θέσης που κατέχουν στην κοινωνία, λόγω του διαφορετικού ποσοστού των ανδρών που εργάζονται και των γυναικών που εργάζονται ή των ανδρών που μένουν στο σπίτι ή των γυναικών που μένουν στο, σπίτι. Πολύ περισσότερες γυναίκες περπατούν και διανύουν πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις για να έχουν πρόσβαση σε νερό ή σε οτιδήποτε άλλο. Και βεβαίω υπάρχει πολύ διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης ή μόρφωσης. Όλοι αυτοί είναι οι λόγοι που θα επηρεάσουν τα δύο φύλλα διαφορετικά οι κλιματικές αλλαγές. Εξού και ε, οι πολιτικές για το μετριασμό της επίπτωσης των κλιματικών αλλαγών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη διάσταση του φύλου. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο τώρα υπάρχουν και εκεί βεβαίως ανισότητες και τις γνωρίζουμε όλοι. Ε, ποσοστό, διαφορετικό ποσοστό απασχόληση στην αγορά εργασίας, μικρότερη αμοιβή για την κατάληψη ίδιων θέσεων απασχόλησης, της ίδιας θέσης, λιγότερες γυναίκες στις θετικές επιστήμες. Όλα αυτά ισχύουν. Ενδεχομένως στην Ευρώπη όλα αυτά δεν μπορούμε να τα εξαλείψουμε μέσω της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή. Μεθαύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει για τη μεταρρύθμιση της κυρίας γεωργικής πολιτικής και σε αυτό το κείμενο δεν θα βρείτε τη διάσταση του φύλου αποτυπωμένη λέξη προς λέξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα της ισότητας των φύλων. Ε, επίσης έγινε λόγος για το ποιος έχει την οικονομική δυνατότητα να πάρει πιο αμάξι. Νομίζω ότι η πολιτική για το κλίμα στην Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες. Διότι εάν προχωρήσουμε ε, και επιτύχουμε τους στόχους μας που έχουμε για το κλίμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έχουμε πολύ καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και επομένως πολύ περισσότερες γυναίκες θα κάνουν την οικολογική επιλογή της χρήσης των μέσων μεταφοράς. Επομένως αυτό θα μπορούσε να μας βοηθήσει να ε, εξαλείψουμε τις ανισότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια πρέπει να πω ότι όταν ε, ας πούμε υπάρχουν πλημμύρες φέτος το καλοκαίρι στην Τία Σουηδία ή στη Βόρεια Πολωνία ή στη Βόρεια Δανία εκεί όντως δεν πλήττονται διαφορετικά οι γυναίκες από ό,τι πλήττονται οι άνδρες. Αυτό όμως δεν ισχύει σε άλλα μέρη του κόσμου. Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταία. Όταν ρωτούνται οι γυναίκες και οι άνδρες σε ποια αντίληψη έχουν για το κλίμα, τα, οι αποτελέσματα και απαντήσει μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικά σε άλλα θέματα, αλλά σε αυτό το θέμα είναι αρκετά παρόμοια και παρεμφερεί τα αποτελέσματα και οι απαντήσεις ε, στις διάφορες έρευνες που γίνονται. Αυτός ο διαχωρισμός λοιπόν είναι πολύ σημαντικός. Επειδή πρέπει να φύγω αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνετε, για αυτή την πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει και να πω ότι το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις που διεξάγουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε και η κατανάλωση και θα τα εξετάσουμε αυτά τα θέματα στο Ρίο Plus 20, στο Ρίο Συν 20, που θα είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε και ευχαριστώ που κάνατε και την παρουσίασή σας. Βεβαίως θα συνεχίσουμε την συνεργασία μας μαζί σας. Vi har lite mer tid kvar när det den här momentet, så jag vill fråga, nu har ju då... Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. jag undrar om det finns Υπάρχουν ερωτήματα ή σχόλια, θέλετε να προσθέσετε κάτι ή πέραν των μελών της Επιτροπής θέλει κάποιος άλλος να θέσει κάποιο ερώτημα. Okay. Okay. In that case we move on and we're going to make some switch here. Ωραία. Άρα προχωρούμε. Eh, Ωραία, προχωρούμε λοιπόν. Αλλάξαμε εμπειρογνώμονες, έχουμε δύο νέα πρόσωπα εδώ. Σας καλωσορίζω. Θα έχετε κι εσείς 15 λεπτά για την παρουσίασή σας. Να καλωσορίσουμε την κυρία Λιάνε Σάλατεκ από το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ της Αμερικής. Ε, μπορείτε να μας συστηθείτε πριν ε, παρουσιάσετε τα όσα έχετε να πείτε. Ευχαριστώ. Καταρχάς ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω σήμερα. Δυστυχώς δεν έχω παρουσίαση PowerPoint και αποφάσισα να μην κάνω τέτοια είδους παρουσίαση γιατί η δική μου παρουσίαση έχει να κάνει με την χρηματοδότηση για το κλίμα. Είναι σημαντικό λοιπόν να επικεντρωθούμε σε κάποιες ε, αρχές και θα ήθελα να παραμείνω σε αυτά. Ο τίτλος λοιπόν της παρουσίασης μου είναι αυτό. Ε, η, το, η χρηματοδότηση του κλίματος, ε, διπλό mainstreaming για την βιώσιμη ανάπτυξη. λόγω και της ε, ε που υπάρχουν μεταξύ των φύλων, των προτύπων, ε, των ε, προβλημάτων που αντιμετωπίζονται σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε πόρους, τη φτώχεια. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στους οικονομικούς πόρους που δεσμεύονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της σε παγκόσμιο επίπεδο για να αντιμετωπιστούν οι κλιματικές αλλαγές ό,τι αφορά την, την προσαρμογή ως προϋπόθεση για να υπάρξει ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών. Όπως ακούσαμε, το, ε, η, σύμβαση πλαίσιο του ΟΗΕ για τις κλιματικές αλλαγές ε, αρχίζει να συμπεριλαμβάνει κάποια διατύπωση, κάποιες αναφορές στα δύο φύλλα. Η Επίτροπος ε, Χέντεγκαρ Καρδιστικός δεν είναι εδώ, αλλά το είπε. Ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια αναφορά στα φύλλα, στην ισότητα των φύλων, ως ένα οριζόντιο διατομιακό θέμα, ακόμη και με ε, οδικούς χάρτες που θα μπορούσαν ίσως να θεωρούνται άσχετοι με αυτό, όπως ας πούμε η πολιτική γεωργία, η ενέργεια, η κλιματική πολιτική κτλ. Το, η σύμβαση λοιπόν πλαίσιο του ΟΗΕ ξεκίνησε με την τελευταία συμφωνία στην Κανκούν να αναγνωρίζει το θέμα της ε, ισότητας των δύο φύλων και της ε, συμμετοχής των γυναικών και βάζει την πτυχή αυτή σε όλες τις πτυχές της, ε, των κλιματικών αλλαγών. Και επίσης επιβεβαιώθηκε, επιβεβαιώθηκαν οι οικονομικοί στόχοι, μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι, για την ε, χρηματοδότηση της, ε, του κλίματος με συμμετοχή όλων των κρατών μελών ώστε να υπάρξει ε, νέα επιπλέον χρηματοδότηση για να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν προβλήματα μέσω της προσαρμογής και της διάσωσης των δασών τους. Ακούσαμε ποιες είναι οι ανάγκες, το είπε και η Επιτροπός, ότι χρειαζόμαστε όντως άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του κλίματος, των κλιματικών αλλαγών. Αυτές οι δράσεις όμως χρειάζεται να ε, συμπεριλαμβάνουν και τα απαραίτητα μέσα που να συμπεριλαμβάνουν την πτυχή των φύλων. Αυτό είναι ένα θέμα αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα χρηματοδότηση για, ε, για τις χρηματικές αλλαγές που αναγνωρίζει ότι οι γυναίκε είναι η πιο μεγάλη ε, συμμετέχουσα ομάδα. Δεν μιλάμε για το 10% του παγκοσμίου πληθυσμού, μιλούμε για το 50 ή 52% του παγκοσμίου πληθυσμού. Η εμπειρία από την χρηματοδότηση, την αναπτυξιακή, εκεί μπορεί να παίξει ρόλο γιατί έχει δείξει ότι η ευαισθητοποίηση ό,τι αφορά τα φύλλα για, το σχεδιασμό των προγραμμάτων βελτιώνει τα αποτελέσματά τους και την αποδοτικότητα της χρηματοδότησης αυτής. Αλλά υπάρχει και θέμα υπαρχουσών υποχρεώσεων δυνάμει των διεθνών, ε, του διεθνούς δικαίου για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι αποφάσεις αυτές για τη χρηματοδότηση για το κλίμα δεν γίνονται μέσα σε ένα νομικό κενό και θα πρέπει μια προσέγγιση να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα για τις κλιματικές αλλαγές και τις σχετικές δράσεις ε, και να μπορεί να λάβει υπόψη της ε, όλα τα, όλες τις πτυχές ε, όπως και το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν και κάποιες παραβιάσεις. Παρ' όλα αυτά, αν δούμε τους μηχανισμούς χρηματοδότησης, γενικώ έχουν αποτύχει ώστε να θεωρήσουν τη γυναίκα έναν βασικό παίκτη συνήθως μιλούμε μόνο για ευαίσθητες ομάδες, το ακούσαμε και ήδη σήμερα το πρωί. Και αυτό βεβαίως δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται σαφέστερη αναγνώριση των φύλων, αντρών και γυναικών. Σήμερα η χρηματοδότηση η δημόσια ε, ακόμα δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη της το θέμα των δύο φύλων και αυτό μπορεί να γίνει μέσω. Ε, αυτό είναι άσχετο μάλλον με το αν η χρηματοδότηση αυτή πάει σε πολυετή ή διμερεί ε, σχέσει ή προγράμματα ε, για την χρηματοδότηση του κλίματο ε, και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών του, όπως ας πούμε το Rio Markers, οι δείκτες του Rio του ΩΣΑ. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για την διεύρυνση των διαπραγματεύσεων για τη χρηματοδότηση και για την ε, ε, σωστή διάδοση των ε, κονδυλίων. Αυτό αναφέρεται και στη UNFCCC και στο G7 και στο G20 που συζητά τώρα ακριβώς τους πόρους αυτής της χρηματοδότησης. Είναι σημαντικό θέμα και για την Παγκόσμια Τράπεζα και για την Τράπεζα Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και την, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις ε, και τις εθνικές ε, τράπεζες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι ένα διπλό mainstreaming. Δηλαδή το mainstreaming της, ε, η συμπερίληψη δηλαδή του κλίματος ε, και στην αναπτυξιακή πολιτική που συμπεριλαμβάνει όμως και μία προσέγγιση mainstreaming για τα φύλλα για να επιτύχουμε τον στόχο που ο στόχος είναι χαμηλό, χαμηλός άνθρακας ε, με ανοχή, οικονομία δηλαδή χαμηλού άνθρακα με, ανοχή στην, στις κλιματικές αλλαγές και ισότητα για τα δύο φύλλα. Όταν λοιπόν ορίσουμε ποιες είναι οι ανάγκες μας θα δούμε ότι υπάρχει σαφές κενό μεταξύ των αναγκών χρηματοδότησης από τις αναπτυσσόμενες χώρε και το, της χρηματοδότησης που τελικά δίνεται από τις, από τις αναπτυσμένες χώρες. Και αυτό οφείλεται στο ότι οι περισσότεροι διμερείς μηχανισμοί χρηματοδότησης βασίζονται κυρίως σε θελοντικές πληρωμές αντί για υποχρεωτική αξιολόγηση ε, προϋπολογισμού των αντιναπτυσσόμενων χωρών και έχετε, ε, δηλαδή υπάρχουν πολλές προσφορές αλλά δεν μεταφράζονται τελικά σε με σε συγκεκριμένη καταβολή κονδυλίων. Επίσης σημαντικό, για την, όπως ε, εξίσου σημαντικό με την ποσότητα, είναι και η ποιότητα για τη χρηματοδότηση του κλίματος. Υπάρχουν κάποιες αρχές που είναι βασικές και που θα πρέπει να εφαρμόζονται για το, σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση. Θα πρέπει να, υπά, να είναι προβλέψιμο ε, το, η εξασφάλιση της ε, μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ε, με βάση τα προγράμματα και θα πρέπει επίσης να βασίζεται στις ε, βασικές ε, ευθύνες. Ας πούμε, ο ρηπαίνων πληρώνει. Ε, θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο νέα και καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης, όπως ο φόρος για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή θα είναι επιπλέον των υπαρχόντων προγραμμάτων των Αυτέ οι ποιοτικέ αρχές λοιπόν και τα κριτήρια για την δημόσια χρηματοδότηση για το κλίμα είναι σημαντικά και βεβαίως σχετικά με το φύλλο. Για παράδειγμα, όταν η, η χρηματοδότηση για την προσαρμογή δίδεται σε φτωχέ χώρες ω ε, δάνεια, συμβάλλει, στις φτωχές χώρες συμβάλλει στο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που, που υπάρχουν στις χώρες αυτές, ε, που βεβαίως συχνά υπάρχουν στον ε, σε ό,τι αφορά την μείωση θέσεων εργασία σε τέτοια κοινωνικά προγράμματα και ε, μια που η χρηματοδότηση αυτή χρησιμοποιεί τα χρήματα των φορολογουμένων, η κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι ε, η διαφάνεια και η ευθύνη, η λογοδοσία και η συμμετοχή ε, είναι εξασφαλισμένες. Η εφαρμογή αυτών των βασικών αρχών είναι προϋπόθεση ώστε η χρηματοδότηση των κλιματικών αλλαγών να είναι πιο ισότιμη όσο αφορά τα φύλλα, να δίδονται στις γυναίκες οι, ε, οι πληροφορίες και η γνώση για να μπορέσουν να συμμετέχουν και να λαμβάνουν αποφάσεις σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Ποιες είναι οι βασικές αρχές και δράσεις. Σίγουρα δεν θα σας τις πω όλες, δεν θα προλάβω. Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό η ισότητα των φύλων αποτελέσει την ε, βασική αρχή ε, σε όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης. Θα πρέπει να αποτελέσει βασική αρχή των, του Παγκοσμίου Ταμείου ε, για την αντιμετώπιση του AIDS, ας πούμε, της εφηματίωσης, της ελονοσίας και του, της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τα, για τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς. Μέχρι στιγμή οι εξελίξει στον τομέα αυτό έχουν γίνει πάρα πολύ, έχουν, είναι πάρα πολύ αργέ. Και έχουμε και το θέμα του retrofitting, το οποίο επίσης πρέπει να σκεφτούμε. Πρέπει να έχουμε σαφείς κατευθυντήριες γραμμέ και κριτήρια για την ε, χρηματοδότηση που πρέπει να είναι συγκεκριμένα για κάθε, ε, για κάθε τομέα. Ας πούμε, ε, όταν υπάρχει θέμα ε, ενδιάμεσης παρέμβασης. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις πιο μικρές κοινότητες, με τις προσπάθειες που γίνονται από χώρες για την μικρότερη εκπομπή αερίων. Θα πρέπει να ε, συγκεντρωθούμε σε συγκεκριμένες κλίμακες. Ας πούμε, η ε, οι κουζίνες, οι ηλεκτρικές κουζίνες, οι συσκευές είναι πάρα πολύ, ε, είναι ένα σημαντικό παράγοντας που πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη μα. Επίσης, κριτήρια ειδικά για τα φύλλα πρέπει να συμπεριληφθούν στα, στα μέσα χρηματοδότηση. Αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένη ανάλυση υποχρεωτική για τα φύλλα για κάθε πρόγραμμα. Θα πρέπει να υπάρχει ε, προπολογισμό για τα φύλλα και θα πρέπει να υπάρχουν και σαφείς δείκτες που θα μετρούν πώς αυτά τα προγράμματα συμβάλλουν στους στόχους για την ισότητα των φύλων. Νομίζω ότι το έχουμε πολλές φορές, αλλά είναι σημαντικό να συλλέγουμε συστηματικά τέτοια δεδομένα που αφορούν τα δύο φύλλα. Να υπάρξουν, ας πούμε, ε, συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία θα τα προχωρούμε, θα τα παρακολουθούμε και θα έχουμε και σαφείς δείκτες για τα δύο φύλλα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα, δεδομένα αυτά για τα φύλλα ε, βρισκόμαστε στην ε, περίπτωση του ε, αν έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Δεν έχουμε επαρκή ε, δεδομένα για να ε, στοιχειοθετήσουμε τα προγράμματα που θέλουμε. Πρέπει λοιπόν να τα συλλέξουμε. Ας ξεκινήσουμε. Ακούσαμε και για το Ευρωβαρόμετρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο μπορούν να αποτελέσουν τους μοχλούς για να ζητήσουμε και για να πιέσουμε για τη συλλογή τέτοιων δεδομένων. Χρειαζόμαστε ε, ισορροπία σε ό,τι αφορά την, ε, τα φύλλα στην λήψη αποφάσεων και χρειαζόμαστε και εμπειρογνωμοσύνη πάλι για τα δύο φύλλα όταν μιλούμε για χρηματοδότηση του κλίματος. Είναι απαραίτητο αυτό γιατί αλλιώς αυτές οι πτυχές της ισότητας των φύλων δεν θα συμπεριλαμβάνονται σε προγράμματα και projects. Χρειάζεται συμβολή και συμμετοχή των, ε, γυναικών ως ενδιαφερομένων μερών και ως ε, επιλέξιμων για χρηματοδότηση. Βεβαίως αυτό στα πλαίσια και των εθνικών ε, προγραμμάτων που υπάρχουν και των προγραμμάτων προσαρμογής. Αλλά θα πρέπει να υπάρξουν ανάλογα με τη χώρα και ανάλογα με το φύλλο τέτοια προγράμματα διαφανή και συγκεκριμένα. Γιατί οι άνθρωποι που θα ε, εποφεληθούν από, από τη χρηματοδότηση αυτή θα είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται επιτόπου τόπου στις χώρες αυτές. Επίσης, γενικός έλεγχος της, ε, ε, της χρηματοδότησης και για την ε, χρηματοδότηση για το κλίμα και για την ανάπτυξη. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το DAC, μόνο 22% της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αφορά, ε, ασχολείται με θέματα ισότητας των δύο φύλων. Mm. Το gender mainstreaming λοιπόν είναι μία από τις βασικές αρχές για την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας. Και λίγο πιο γρήγορα, ε, κάποια βασικά πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο μεγαλύτερος ε, πάροχος τέτοιας χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και για το κλίμα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 27 κράτη-μέλη της έχουν ειδική ευθύνη να δράσουν ως βασικοί ε, παίκτες στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης με βάση το φύλλο για το κλίμα. Επίσης, για το, έχουμε το, την ε, σύνοδο στο Ντερμπάν για την, του COP17 για το, για το Πράσινο Ταμείο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, θέσει το θέμα της ε, ύπαρξης της πτυχής των φύλων. Και τέλος, και αλήθεια είναι το τελευταίο μου σημείο, το Κοινοβούλιο ε, που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους ε, πολίτες έχει ειδική ευθύνη να ε, ζητήσει την λογοδοσία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο δαπανά τα χρήματα των φορολογουμένων. Θα πρέπει να ζητήσει ε, η χρηματοδότηση για, την, ε, για το κλίμα και την ανάπτυξη να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της, των, περιφερειακών, των ε, γειτονικών χωρών και, και σε όλο τον κόσμο, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα και ανοχή στο κλίμα. Αυτό συμπεριλαμβάνει και δράσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και τα κονδύλια που ήδη δίνονται από, το, από τη Συμμαχία για την αλλαγή του κλίματος και, την, και το Ταμείο για την ενεργειακή απόδοση και τις ε, ανανεώσιμες ε, ενέργειες, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνουν αυτή τη στιγμή την πτυχή των δύο φύλων. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε, είπατε. Som ναι, βεβαίως ε, είναι πολύ σημαντικό το συμπέρασμα το οποίο καταλήξατε. Και ε, φυσικά η ισότητα των φύλων θα πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη σε όλα τα οικονομικά και χρηματοδοτικά ζητήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σαλατέκ. Ε, Alder θα παρουσιάσει τον εαυτό σου πριν κάνεις ε, την παρουσίαση, έτσι, ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για αυτήν την ακρόαση την οποία περιμέναμε καιρό. Εμείς ε, δουλεύουμε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ε, για το θέμα γυναίκες και κλιματικές αλλαγές. Κυρίως εδώ ε, ξεκινήσαμε από τις χώρες Αφρικής και τον αναπτυσσόμενο κόσμο και είναι εξαιρετικό τώρα το ότι μας απασχολεί και στην Ευρώπη πλέον. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα προχωρήσει, θα διευρυνθεί η συζήτηση. Ίσως πρέπει να σας εξηγήσω δύο-τρία πράγματα γιατί ενδεχομένως Ε, δεν γνωρίζετε τη διαδικασία UNFCC. Ε, το UNFCC, η διαδικασία UNFCC σημαίνει ότι ορισμένες ε, χώρες μέλη ε, παρακολουθούν τις, ε, και διεάγουν μάλλον τις συζητήσεις αλλά υπάρχουν και, μην, και, και κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις συγκεκριμένα 1.500 είναι αυτές οι οργανώσεις οι οποίες παρακολουθούν από κοντά τις συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή. Ε, εμείς είμαστε ε, περίπου 6-7 μικρές ε, οργανώσεις. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας δώσω την διάσταση των γυναικών στη διαδικασία UNFCC Ε, η αντιμετώπιση που έχουμε είναι δυτή, δηλαδή πρώτα απ' όλα ε, ε, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και δεύτερον προσαρμογή ε, στην διαδικασία στη συμφωνία του Κανκούν υπάρχει μια της Κανκούν μάλλον υπάρχει μία αναφορά στην ισότητα των φύλων αλλά σπανίζει γενικώ όσον αφορά την προσαρμογή. Ε, όσον αφορά τώρα τον μετριασμό των ε, αποτελεσμάτων εκεί και σε διεθνές επίπεδο ε, γίνεται, γίνεται αναγνώριση του, της παρουσίας ε, των ε, αναπτυσσόμενων χωρών ε, στο, στα θέματα αυτά, εκτός από τα θέματα της, των δασών και της υλοτομίας. Επίσης υπάρχει κάποια αναφορά γλωσσική στις διατυπώσεις στην ισότητα των φύλων στο πρωτόκολλο της Κανκούνα, αλλά η κύρια δεσμευτική συμφωνία ε, σχετικά με τον μετριασμό των επιπτώσεων ε, η πρώτη περίοδος έντροφης οργανών το 2012 και επομένως θα δούμε μετά τι θα γίνει και ε, ποιε θα είναι οι μελλοντικές δεσμεύσεις οι οποίες θα αναλυφθούν Επόμενο σημαντικό σημείο είναι η χρηματοδότηση. Πολλά ακούσαμε ε, για την ε, χρηματοδότηση. Επίσης, ε, τεχνολογία. Ήθιστε να λέμε μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Εμάς, εμείς προτιμούμε την έκφραση ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Και πιστεύουμε ότι όλη αυτή η μεταφορά τεχνολογίας έχει να κάνει και με την ισότητα των φύλων. Δηλαδή, τι είδους τεχνογνωσία και τι ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Ε, ε, η, η οικοδόμηση ικανοτήτων, βεβαίως και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα συζητηθεί ε, στην Durban, στο και υπήρχε μια πρώτη αναφορά στη Συμφωνία της Κανκούνα Οι μεγάλες προκλήσεις πάντως βρίσκονται στον μετριασμό. Κατά την άποψή μου και κατά την άποψή μας πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση όσον αφορά την ισότητα των φύλων και στις αναπτυσσόμενες και στις αναπτυσσμένες ε, χώρες. Γιατί η κοινωνία με χαμηλή εκπομπή διοξιδίου του ε, άνθρακα ε, σημαίνει κοινωνία η οποία αλλάζει τις συνήθειές της ε, και για τις ε, βιομηχανικές ε, χώρες, για τις αναπτυγμένες χώρες, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και τώρα που ξέρουμε τόσα πράγματα, ξέρουμε ότι θα πρέπει να μειώσουμε κατά 80% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό σημαίνει μεγάλη αλλαγή στις τεχνολογίες, μεγάλη αλλαγή στον τρόπο ανάπτυξης που έχουμε ακολουθήσει. Με αυτό συνδέεται κάτι που έχει ήδη αναφερθεί από την Ιωάννα. Δηλαδή αυτό που χρειαζόμαστε είναι ε, αναγνώριση της διαφορετικότητας ε, στο θέμα ε, του ίχνους άνθρακα των τροφίμων οι διατροφικές συνήθειες μεταξύ άνδρων και γυναικών διαφέρουν. Οι διατροφικές συνήθειες μεταξύ αναπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου επίσης ε, διαφέρει. Οι προτιμήσεις είναι διαφορετικές. Επομένω, ποιες πολιτικές επιθυμούν να δουν οι γυναίκες, ποιες είναι οι πολιτικές που οι άνδρες επιθυμούν να δουν. Ε, αυτό το αναφέρω κυρίως στο επόμενο σημείο μου, δηλαδή στο lifestyle, στον τρόπο ζωής στις ε, διεθνείς ε, διαπραγματεύσεις για το κλίμα ε, έγινε μεγάλη εστίαση στην οικονομία και την τεχνολογία. Κανείς όμως δεν αναφέρθηκε στις δομές, στις υποδομές, την υποδομή των δημοσίων μεταφορών και βεβαίως και τον τρόπο ζωής, το lifestyle. Από συγκεκριμένες μελέτες που έχουν γίνει σε ολόκληρο τον κόσμο, κυρίως στην Ευρώπη, γνωρίζουμε ότι εάν ε, ε, ε, θέσει κανείς το ερώτημα των προτιμήσεων, οι άνδρες θα προτιμήσουν μεγαλύτερη επένδυση στην τεχνολογία, ενώ οι γυναίκες θέλουν αλλαγή των δομών και του τρόπου ζωής. Οι γυναίκες λοιπόν πιστεύω ότι θα έδιναν καλύτερες, καλύτερες θέσεις και αν αυτές έλαβαν τις αποφάσεις τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα όσον αφορά την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών έτσι ώστε να βελτιώσουμε τη θέση των φύλων. Νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει απλά η διατύπωση στα κείμενα γιατί έχουν γίνει, έχουν γίνει κάποιες μελέτες, έχει εισαχθεί η λεγόμενη gender language ε, στα, ε, στα κείμενα. και έτσι όπως βλέπω εγώ τα πράγματα ε, νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερες ε, ε, μεγάλες λύσεις παρά σωστές λύσεις. Υπάρχουν πολλές χώρες που θέλουν την βιομηχανική. Είναι πολλοί αυτοί που δεν θέλουν πλέον την πυρηνική ενέργεια ε, γίνεται πλέον λόγος ε, για τους ωκεανούς or for instance plantations um, with genetically modified organisms και την ε, καλλιέργεια στο πούμε των ωκεανών θέματα τα οποία δεν γίνονται δεκτά από την ε, πλειοψηφία των, ε, ε, γυναικών αλλά αυτές οι ψεύτικες λύσεις μάλλον κερδίζουν έδαφος Επίσης, στα πλαίσια των διεθνών εξελίξεων και διαπραγματεύσεων θα πρέπει να υπάρχει ε, κάποια εκπροσώπηση καλύτερη των γυναικών γιατί ε, δεν υπάρχει αρκετή τεχνο, αρκετή πραγματογνωμοσύνη όσον αφορά ε, τις, τα θέματα των γυναικών. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Όσον αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπω τρεις ε, μεγάλους, ε, μεγάλους τομείς ε, στους οποίους μπορεί να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει προενεργητικό ρόλο όσον αφορά πιο φιλόδοξες πιο φιλόδοξες απαιτήσει. Είναι γεγονό ότι πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη επίσης θα πρέπει να ε, είναι πρωτοπόρος όσον αφορά την, ε, τη θέση των γυναικών και τη θέση των δύο φίλων όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Ε, στην ε, Φιλανδία είδαμε ότι ε, έχουν μόνο γυναίκες στην αντιπροσωπεία τους έτσι ώστε να υπάρξει μια εξισορρόπηση με τις χώρες οι οποίες δεν έχουν σημαντική εκπροσώπηση γυναικών αλλά βεβαίως πρέπει να υπάρχει εξισορρόπηση και το σημαντικό είναι να μιλάει η Ευρώπη με μία, με μία φωνή. Ε, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη διάσταση όσον αφορά και πολλές ε, ελλείψεις όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών αλλά παρόλα αυτά πολλά γίνονται και βεβαίως ε, σε επίπεδο κεντρικών αποφάσεων αλλά νομίζω ότι πολλά μπορούν να γίνουν και στην κάθε χώρα ξεχωριστά και σε πιο χαμηλό επίπεδο. και νομίζω ότι θα πρέπει ε, και στη διαδικασία μετριασμού και στη διαδικασία προσαρμογής να ε, βρουν οι γυναίκες τη θέση τους, ε, κυρίως όσον αφορά τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Αυτά τα λίγα για να σας θυμίσω λίγο ή να, το, επανατοποθετήσω τις γυναίκες στον γενικότερο, στην γενικότερη εικόνα. Ε, first, power η συμμετοχή στη διαδικασία λήψεων αποφάσεων ε, πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί στην ουσία μιλάμε για ενεργειακή πολιτική, μιλάμε για, ε, για πολιτική μεταφορών και βλέπετε στις εικόνες πώς παρουσιάζονται τα πράγματα. Κάτι άλλο που ε, αναφέρθηκε προηγουμένως η διαφορά ε, στις αμοιβέ ε, που βεβαίως κάνουν τις γυναίκες πιο ευάλωτες αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την οικονομία της φροντίδας. Γνωρίζουμε ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της μη αμοιβόμενη ε, ε, παροχής ε, φροντίδας. Υπάρχουν διαφάνειες γι' αυτό. Εδώ βλέπετε και φωτογραφίες από την Γερμανική Επιτροπή Ενέργειας που οθούν τους ανθρώπους να καταναλώσουν πιο σωστά την ενέργεια. Πολλά μπορούν να γίνουν λοιπόν. Ε, και ε, There are still also the gender identities, whether we want them or not. That, that... Ε, και ο, ο καθένας ε, πραγματικά θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του με τα μέσα που έχει στη διάθεσή του. To, to suggest or recommend Of Βεβαίως χρειαζόμαστε την αποτελεσματική συμμετοχή των γυναικών και βεβαίως θα πρέπει να ξεπεράσουμε ε, την, ε, αυτό το παιχνίδι των αριθμών στο οποίο συνήθως εξαντλείται η ισότητα των φύλων. Γιατί να ε, μην θεωρηθεί η ισότητα των φύλων σαν, μία, σαν ένας από τους στόχους κεντρικής πολιτικής Ας πούμε στην Σουηδία ε, πέρσι είχαν κύριο στόχο της ε, πολιτικής μεταφορών την ισότητα των φύλων. γιατί είδαν ότι χωρίς ισότητα φύλων και στον τομέα αυτό δεν θα, θα, υπήρξε, ε, θα υπήρχε αύξηση των διακρίσεων κτλ. Θεσμική αντιμετώπιση λοιπόν. Αυτό είναι ένα μεγάλο διακύβευμα και επομένως όλοι ε, αυτοί που είναι υπεύθυνοι για, τις, ε, για, το, για τις, την ισότητα των φύλων και αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την κλιματική αλλαγή θεσμικά να συζητήσουν, να επικοινωνούν οι μεν με τους δε. Γιατί ε, αυτό που μάθαμε από τα διεθνή φόρα είναι ότι οι, αυτοί που ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή και αυτοί που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων μιλούν δύο τελείως διαφορετικές γλώσσες. Πρέπει να μάθουν να μιλάνε μεταξύ τους. Και βεβαίως θα πρέπει να εξευρεθεί μια ε, σωστή ένα, να βρεθεί ένα σωστό θεσμικό πλαίσιο ε, έτσι ώστε να συζητούν μεταξύ τους ας πούμε οι επιτροπές μεταφορών, οι επιτροπές ενέργειας και ε, αυτοί που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων. άλλο σημείο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό από την πλευρά ε, της ισότητας των φίλων αλλά και από την πλευρά της δικαιοσύνης θα έλεγα εγώ. αυτό που χρειαζόμαστε όταν, μιλάμε για κλιματική αλλαγή δεν είναι να μειωθούν μονάχα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Πρέπει να έχουμε πιο μακρόθωρη πολιτική, θα πρέπει να είναι πιο μακρόπνοα τα σχέδιά μας. Θέλουμε βεβαίως ε, θέλουμε βεβαίως μια κοινωνία η οποία θα καταναλώνει, θα έχει μικρό, ε, χαμηλές εκπομπές ε, άνθρακα, αλλά θα θέλουμε, και μια κοινωνία η οποία θα είναι πιο ανθεκτική από κάθε άποψη. Και βεβαίως να, να ξεπεράσουμε την τυφλότητα όσον αφορά ε, την ισότητα των φύλων αλλά και την κοφότητα όσον αφορά την, τον, τον, ε, την, ισότητα των φύλων. We need, of course, Χρειαζόμαστε όμως και ερμηνείες. Ε, καλό είναι δηλαδή να έχουμε τα αριθμητικά στοιχεία, αλλά χρειαζόμαστε και ερμηνείες, εξηγήσει των στοιχείων αυτών, έτσι ώστε να εξηγούνται όλες αυτές οι διαφορές. Ε, για όλα τα θέματα συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς άνθρακα από την πλευρά των γυναικών, ας πούμε, ήταν προβληματικό ότι ο μηχανισμός ο μηχανισμός αυτών των πόντων ε, και του εμπορίου ε, άνθρακα μας δημιουργούσε πρόβλημα. Γιατί στην ουσία εμποδίζει ε, μάλλον παροτρύνει ανάπτυξη προγραμμάτων τα οποία ούτε κοινωνικά ούτε περιβαλλοντικά είναι σωστά. Και βεβαίως ε, πρέπει να δούμε και τον αντίκτυπο των πολιτικών που αναλαμβάνουμε εδώ στην Ευρώπη. Χαίρομαι πραγματικά που το Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων ε, έκανε αυτήν την μελέτη, της οποίας είμαι μία εκ των ε, ε, συγγραφέων και ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα χρησιμοποιήσει τη μελέτη αυτή. Επίσης πρέπει να δούμε από πιο κοντά τον ρόλο των γυναικών αλλά και τον ρόλο των ανδρών όσον αφορά ε, την προσαρμογή. Γιατί αν δούμε μόνο τον ρόλο των γυναικών θα διαπιστώσουμε ότι οι γυναίκες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αισθάνονται μεγαλύτερη, αυξημένη ευθύνη για το περιβάλλον. Έχουν όλο και περισσότερη διάθεση και βούληση να κάνουν κάτι, να κάνουν τον κόσμο καλύτερο και να κάνουν προσπάθειες όλο και πιο αποτελεσματικές. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι κάνουν και οι άνδρες. Οι άνδρες που εξακολουθούν να οδηγούν μεγάλα αυτοκίνητα. Θα πρέπει να βρούμε, εν πάση περιπτώσει, το σωστό τρόπο ε, και τα κατάλληλα, τις κατάλληλες πολιτικές έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κάνατε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τη σημείωσα και παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας γενικότερα. Πιστεύω ότι τηρείτε τη διάσταση του φίλου και στην πολιτική αυτή αλλά και στις υπόλοιπες. Και εμείς είμαστε αυτής της άποψης. Είναι αδύρυτη ανάγκη να εφαρμόζεται και να ενσωματώνεται η διάσταση του φύλου σε όλους τους τομείς. Έχουμε τις δύο σκιώδες εισηγήτριες. Θα τους δώσω το λόγο, αλλά καταρχάς να δώσω το λόγο στην κυρία Κιλ Νίλσεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρουσιάσω κάποια παραδείγματα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να πείσουν αυτούς που δεν βλέπουν ε, τη σύνδεση μεταξύ ε, γυναικών διάστασης του φύλου και κλιματικής αλλαγής. Η κυρία Γιανακουδάκη δεν είναι εδώ, αλλά θα τη δω αργότερα και θα το συζητήσω μαζί, σας, μαζί της. Το 1998 με τον ε, τυφώνα Μίτς μόνο σε μία πόλη στις Ονδούρες δεν είχαμε κανένα θάνατο λόγω χάρη ε, σε ένα σύστημα προειδοποίησης που είχαν θεσμοθετήσει οι γυναίκες του χωριού και στην Τανζανία. Μία μη κυβερνητική οργάνωση είχε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για να ε, γίνει ένα πηγάδι σε ένα χωριό και μέσα σε δύο χρόνια είχε αποξηρανθεί το πηγάδι γιατί η συζήτηση και προγραμματισμός είχε γίνει μόνο με τους άνδρες του χωριού. Στη συνέχεια οι γυναίκες που αυτές πήγαιναν να ε, αντλήσουν το νερό ήξεραν στο παρελθόν που ε, αναζητούσαν το νερό και από πού το αντλούσαν. Το αντλούσαν από διαφορετική τοποθεσία από αυτήν στην οποία είχε ε, χαραχθεί το είχε σχεδιαστεί να γίνει το πηγάδι. Επομένως, αν είχε γίνει εκεί, δεν θα είχε εξεραθεί μέσα σε δύο χρόνια. Και έχουμε και τα παραδείγματα της ε, φύτευσης δασών στην Αφρική. Αλλά και αλλού. Στο Ελσίνκι, αν δεν απατώμε, για να περάσουμε και ε, στα ευρωπαϊκά πράγματα, έγιναν συναντήσεις με γυναίκες για να αποφασιστεί ότι τα λεωφορεία οφείλουν το βράδυ να σταματήσουν όχι μόνο στις στάσεις αλλά μεταξύ των στάσεων διότι μπορεί να υπήρξε πρόβλημα ασφάλειας. Δηλαδή, μια γυναίκα που γυρνούσε με το λεωφορείο το βράδυ στο σπίτι της μπορούσε να ζητήσει από τον οδηγό να μην σταματήσει στη στάση αλλά να σταματήσει στο κοντινότερο σημείο της διαδρομής ε, στο κοντινότερο σημείο ως προς το σπίτι της έστω και αν δεν ήταν ακριβώς η στάση αυτή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης δωρεάν μεταφορά ε, για οποιονδήποτε κυκλοφορεί με καροτσάκι, με μωρό μέσα. Είτε είναι γυναίκα είτε είναι άνδρες. άνδρας. Όλες αυτές ήταν συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν από γυναίκες και είναι Αυτά τα συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, γι' αυτό και ζήτησα το λόγο κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος και εγώ ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Σύρπα Πιετικάινεν, σκιώδη εισηγήτρια για το ΕΛΚ. Πέντε λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που δεν απαρέστην στη συνεδρίαση από την έναρξη της. Η βοηθός μου ήταν εδώ, εγώ είχα λιμένες υποχρεώσεις και έχει κρατήσει σημειώσεις και βεβαίως θα ενημερωθώ για όλα ε, τα αποτελέσματα. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες της κλιματικής αλλαγής. Όλοι γνωρίζουμε τις προκλήσεις που υψώνονται μπροστά μας. Ένα σημείο θέλω να υπογραμμίσω, ότι χρειαζόμαστε μια συστημική και συστηματική προσέγγιση Δηλαδή να μην έχουμε μία ε, προσέγγιση μίας γνώμης μόνο, μίας οπτικής γωνίας. Το ποσοστό του 80% είναι πολύ σημαντικό. Εγώ ήμουν μία από αυτές που το υποστήριζαν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δεσμεύσουμε ακόμα περισσότερο ε, διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, από αυτό που είχαμε σχεδιάσει εξ αρχής. Πρέπει να φτάσουμε στο 100%. Αυτό φαίνεται πλέον ξεκάθαρα. Ωστόσο, ε, η συστημική προσέγγιση απαιτεί ε, την εμπλοκή των γυναικών. Καταρχάς, ο αντίκτυπος και δεύτερον η δράση. Αντίκτυπος θα είναι η ενσυναίσθηση ότι οι γυναίκες είναι η ομάδα που θα υποφέρει περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. Και βεβαίως οι αυτόχθονες πληθυσμοί, οι ηθαγενείς, οι φτωχοί, και ούτω καθεξής θα είναι αυτοί που θα υποφέρουν περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες απανταχού στη γη και υπερεκπροσωπούνται στα αριθμητικά στοιχεία που μετρούν τη φτώχεια. Υπερεκπροσωπούνται ως άτομα που εξαρτώνται από άλλους ή που διαβιώνουν σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Το γεγονός λοιπόν παραμένει όταν η κλιματική αλλαγή ε, φτάσει στο απόγειό της θα πλήξει περισσότερο την πιο ευπαθή κοινωνική ομάδα, άρα τις γυναίκες μεταξύ άλλων. Και υπ' αυτή την έννοια οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με τη διάσταση των δύο φύλων, είναι ένα θέμα που έχει να κάνει ε, με την ισότητα ανδρών και γυναικών, δεν είναι ένα θέμα η ε, ισότητα ανδρών και γυναικών άσχετο με την ε, κλιματική αλλαγή. Και βεβαίως προτιμώ εγώ ε, να συζητούμε για την ποιότητα και την ισότητα. Οι γυναίκες είναι ο μισός πληθυσμός της γης όχι, μάλιστα με διορθώνετε τώρα, δεν είναι ο είναι 53%, λίγο περισσότερες. Ωστόσο, υποεκπροσωπούμαστε στις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή, όπως και στις άλλες διεθνείς διαπραγματεύσεις. και υπερεκπροσωπούνται βεβαίως στις διαπραγματεύσεις αυτές οι ομάδες που έχουν οικονομικά συμφέροντα. Έχουμε υπερεκπροσώπηση όλων όσοι δεν θέλουν να ληφθούν οι αποφάσεις γιατί θα πληγούν τα οικονομικά του συμφέροντα και υποεκπροσώπηση, υποεκπροσώπηση δική μας με την ιδιότητά μας των γυναικών. Επομένως χρειάζεται ένα κάποιο ε, θεσμικό πλαίσιο ή ένα θεσμικό εργαλείο για να δοθεί περισσότερη δύναμη, περισσότερη ισχύ στις γυναίκες, στις ομάδες γενικότερα που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ή λήψης των αποφάσεων. Και η ανάγκη, η τεκμηρίωση για την ύπαρξη αυτού του θεσμικού πλαισίου είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι αυτές που θα πληγούν περισσότερο. Άρα ε, θα πρέπει να εκπροσωπούνται κατά 50% τουλάχιστον στις διαπραγματεύσεις. Και ένα άλλο θέμα είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων ανατομέα. Όταν π.χ. έχουμε Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας, μπορεί να έχουμε περισσότερες γυναίκες εκεί, αλλά σε Σύνοδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων ή σε Συμβούλιο Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, εκεί σπάνια βλέπουμε γυναίκες, ενώ εκεί αποφασίζονται εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα. Ποια είναι λοιπόν τα νομοθετικά εργαλεία, οι νομοθετικοί μηχανισμοί, οι θεσμικές ρυθμίσεις που μπορούμε να υιοθετήσουμε για να ενισχύσουμε ενισχύσουμε την συμμετοχή. Είναι η αρχή της ισότητας. Οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούνται στο τραπέζι ε, γύρω από το οποίο κάθονται αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Από εκεί και πέρα, μέρος της δράσης μας θα πρέπει να είναι η γνώση. Και αυτό είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με την ποιότητα. Διστάζω λίγο να αναφερθώ στις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών ε, κατηγοριοποιώντας αυτές σε κουτάκια. Αληθεύει το γεγονός ότι έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα στον τομέα της γνώσης ε, τα δύο φύλλα. Αυτό όμω έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν το σύστημα και θα πρέπει να δούμε πώς κατανέμουμε τους πόρους μας. Πάντοτε με εντυπωσίαζε το ενδεχόμενο να βάλουμε στο ίδιο καλάθι τους δείκτες. Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος και ο αντίκτυπος ας πούμε στην ισότητα των φύλων. Να τα εξαρτάσουμε μαζί. Στην περίπτωση των μέσων μαζικής μεταφοράς και, των, ε, ε και της χρήσης ε, ιδιωτικού αυτοκινήτου. Πού είναι καλύτερα να ζούμε, εκεί όπου υπάρχει άμεση πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή εκεί όπου είναι πιο εύκολο να κάνει κανείς ποδήλατο ή ποιο από τα δύο ε, διασφαλίζει περισσότερη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και ποιο από τα δύο διασφαλίζει μια πιο βιώσιμη χρήση των ε, πόρων. Εάν εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα, βλέπουμε ότι πολύ συχνά αλληλοσυνδέονται. Δημιουργείται ένα καλύτερο περιβάλλον και για τα παιδιά, όταν έχουμε πρόσβαση σε υπηρεσίες στην εγκύτερη περιοχή. Ε, βελτιώνουμε την, ε, τον, την κατάσταση ως προς την κλιματική αλλαγή. Αυξάνονται και βελτιώνονται οι προοπτικές. Άρα υπάρχει και μεγαλύτερη ισορροπία ε, στη διάσταση των δύο φύλων. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό όλους τους δείκτες να τους χρησιμοποιούμε μαζί και να τονίζουμε τη γνώση των γυναικών ως προς αυτά. Και αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε ε, ε, και στο σχεδιασμό που θα κάνουμε ε, σε επίπεδο κοινωνίας. Θα μπορούσα να μακρηγορήσω πάρα πολύ για όλα αυτά τα case studies, για όλες αυτές τις περιπτωσιολογικές μελέτες που έχουμε κάνει, οι οποίες μας μαθαίνουν πολλά πράγματα. Πολύ συχνά δημιουργούμε πρόβλημα, ενώ ε, θα έπρεπε να επιμείνουμε ε, στην πιο απλή κλίμακα, στην πιο μικρή κλίμακα και στις πιο απλές λύσεις, γιατί πολύ συχνά είναι αυτές που είναι πιο αποτελεσματικές. Και κατά τρίτο λόγο, νομίζω ότι δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του κλίματος και του περιβάλλοντος γενικότερα χωρίς να έχουμε μια πολύ μεγάλη ε, κοινωνική διάσταση παρούσα εκεί. Ε, αν ε, αυξήσουμε τις ανισότητες θα έχουμε τεράστιες μάχες για το ποιος θα πάρει ό,τι απομείνει. Ενώ αν επιτύχουμε την ισότητα θα φτιάξουμε μια κοινωνία στην οποία να μπορέσουμε να ζήσουμε όλοι. Και κύριε Πρόεδρε, μια τελευταία παρατήρηση. Οι γυναίκες είναι παράγοντες δράσης από τη στιγμή που είναι καταναλώτριες από τη στιγμή που συμμετέχουν και είναι ψηφοφόροι σε μεγάλες πολιτικές δυνάμεις. Θα είμαστε πολύ παραγωγικοί εάν ξεκινήσουμε τέτοιου είδους εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ζητήσουμε στήριξη για γυναικείες οργανώσεις και για άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ούτως ώστε να ευξηθεί η συνειδητοποίηση των γυναικών για όλα αυτά τα θέματα και ούτως ώστε να ενθαρρυνθούν να αναλάβουν δράση σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Μπρίτα Τόμσον, σκιώδη εισηγήτρια των, ε, της προοδευτικής ε, συμμαχίας για των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη γιατί καθυστέρησα και εγώ, διότι είμαι εισηγήτρια για την οδηγία που έχει να κάνει με την ενεργειακή αποδοτικότητα και οφείλω να παρίσταμε σε διάφορες συνεδριάσεις και σε διάφορες αίθουσες ταυτόχρονα. Όταν συζητούμε ε, για την ενέργεια, ε, κάτι το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μέσα στην, στην αίθουσα είναι κυρίως άνδρες, ενώ οι γυναίκες είναι πολύ μεγάλες καταναλώτριες. Και πολύ λίγες γυναίκες επίσης ε, ε, είναι εκεί από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες, εκτός ίσως από τους πρασίνους. άκουσα αυτά που είπατε για τις γυναίκες ως θύματα. Είναι θύματα. Είναι μεν παράγοντες δράσης, αλλά δεν πρέπει να το αρνούμαστε. Ότι είναι θύματα, είναι θύματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Στη Δύση, τουλάχιστον στη δική μου χώρα, Γίνεται πολλή λόγο γι' αυτό ότι πρέπει να σταματήσουν οι γυναίκε να παραπονιούνται και να σταματήσουν να θυματοποιούνται. Εγώ δεν συμφωνώ γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν συγκεκριμένε δομέ στην κοινωνία που θυματοποιούν τη γυναίκα. Πέραν αυτού, στι αναπτυσσόμενε χώρε οι γυναίκες είναι θύματα, είναι σε πάρα πολύ ευπαθή κατάσταση, κυρίως λόγω της φτώχειας. Και ξέρουμε ότι η πλειονότητα των φτωχών είναι γυναίκες. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι γυναίκες πλήττονται πολύ περισσότερο από την κλιματική αλλαγή από ότι οι άνδρες. Το 2012, πότε ήτανε στην Κοπενχάκη, το 2010, με συγχωρείτε λέει ο Μιλήτρια, Είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση ε, που είχε να κάνει με τις γυναίκες στη κλιματική αλλαγή. στην Κοπενχάγη λοιπόν, εκεί ακούσαμε πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες από γυναίκες από όλες τις γωνιές του κόσμου σχεδόν, από τον Μπαγκλαντές, από χώρες της Νοτιοαμερικής, από τον Εμπαπάλ, την Ινδία. Και αυτό που φάνηκε ξεκάθαρα από όλη αυτή τη συζήτηση είναι το εξής. Από τη στιγμή που οι γυναίκες εξαρτώνται από την γεωργική παραγωγή για την επιβίωσή τους, πλήττονται περισσότερο από ό,τι, τους, από ότι οι άνδρες, γιατί οι άνδρες μπορούν να μετακομίσουν και να μεταναστεύσουν στις πόλεις, ενώ οι γυναίκες καλλιεργούν την γη στην Ήπεθρο. Και γι' αυτό είναι εκείνες που πλήττονται περισσότερο από την ε, κλιματική αλλαγή και είναι εκείνες που πλήττονται πρώτες κιόλας θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες ε, μπορούν να μετατραπούν και σε παράγοντες δράσης και αντίδρασης. Πάμε στην Αφρική και βλέπουμε παιδιά, δηλαδή αγόρια, να παίζουν στο νερό και να κολυμπούν και να περνάνε πολύ ωραία. Και τους βλέπει κανείς ε, και λέει πόσο ευτυχισμένα είναι αυτά τα παιδιά παρόλο που είναι φτωχά. Τα κορίτσια όμως δεν είναι έξω και δεν παίζουν με το νερό στη λίμνη ή στο ποτάμι και ως αποτε... το αποτέλεσμα είναι ότι οι γυναίκες δεν ξέρουν να κολυμπούν. Δεν ξέρουν να κολυμπούν γιατί ποτέ δεν έμαθαν να κολυμπούν και γι' αυτό πιο συχνά βρίσκουν το θάνατο ε, σε επόμενη μελλοντική φυσική καταστροφή. Αυτό έγινε με το τσουνάμι στην Ταϊλάνδη. Οι πολλές γυναίκες, οι περισσότερες δεν ήξεραν να κολυμπούν γι' αυτό και το 70% των θυμάτων ήταν γυναίκες σε μια φυσική καταστροφή που έπληξε όλους. Και βέβαια είναι πολύ λίγες οι γυναίκες που παίρνουν μέρος στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Στη χώρα μου, στη Δανία, πηγαίνω σε συνέδρια και οργανώνεται ένα πάρτι το βράδυ και μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο να είμαι σε μια βραδινή εκδήλωση μετά το πρωινό συνέδριο με π.χ. 1500 άνδρες και 30 ε, γυναίκες. Και πρόσφατα πήγα σε ένα άλλο συνέδριο στην Αθήνα με 400 άνδρες και 30 γυναίκες. Στις διαδικασίες και στα φόρουμ που λαμβάνονται ε, αποφάσεις, ε, οι γυναίκες δεν είναι παρούσες. Είναι βασικό θέμα το πώς θα βελτιώσουμε τη συμμετοχή γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Με προσκάλεσαν στην Κίνα πρόσφατα διότι η οργάνωση γυναικών ε, στην Κίνα ε, διοργανώνει ένα συνέδριο για τις γυναίκες και την αηφορία. Θα έχουν εργαστήρια για τις γυναίκες και το κλίμα και ε, προετοιμάζουν μια πολύ μεγάλη κινέζικη αντιπροσωπεία γυναικών η οποία θα παραστεί στις εργασίες του Ρίο Συν 20. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε αντιπροσωπεία για το Ρίο. Μπορούμε να έχουμε, αλλά δεν έχουμε συζητήσει για την εκπροσώπηση των δύο φύλων στην επίσημη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν να το ξεκινήσουμε αυτό, να το κάνουμε, να κάνουμε αυτό το mainstreaming ε, που θα εντάξει τις γυναίκες στη διάσταση του φίλου στην προσπάθεια για περισσότερη αηφορία. Οφείλουμε να αναλάβουμε δράση οφείλουμε να εμπλέξουμε περισσότερο τις γυναίκες ε, στη διαχείριση οικοσυστημάτων σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Να τους δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες στον έλεγχο της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, να διασφαλίσουμε την πρόσβαση των γυναικών στις χρήσεις γης και σε άλλους πόρους. Και βεβαίως να τις εμπλέξουμε στην ε, διαδικασία λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων. Να πω και κάποια θετικά. Τρεις γυναίκες από αναπτυσσόμενες χώρες μόλις έλαβαν τον Νόμπελ Ειρήνης. Και το επιχείρημα ήταν το ακόλουθο. Δεν μπορούμε να πετύχουμε δημοκρατία και μακροημερεύουσα ειρήνη στον κόσμο εάν δεν δοθούν οι ίδιες ευκαιρίες στις γυναίκες όπως και στους άνδρες να επηρεάσουν με τη σκέψη τους ε, τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και εγώ πιστεύω ότι μπορούν να παίξουν μεγάλο ρόλο στην επίτευξη της αηφόρου ανάπτυξης. Γι' αυτό και θα πρέπει να συμμετέχουν και να συμπεριλαμβάνονται σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Ε, και εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην εκπρόσωπο Ροσάριο Μπέντο Παΐς, επικεφαλής του Τμήματος για την Προσαρμογή, Γενική Διεύθυνση για την Κλιματική Αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με καλέσατε να σχολιάσω και να εκφράσω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ είμαι παρούσα από την αρχή της συνεδρίασής μας και επειδή μου ζητήθηκε να σχολιάσω όλες τις παρεμβάσεις, να πω ότι θα σχολιάσω τόσο την πρώτη συνεδρία όσο και τη δεύτερη και έτσι επιγραμματικά ε, θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τι κάνουμε εμείς εδώ. Ακούσαμε λοιπόν ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι ουδέτερη έναντι της ισότητας των φύλων. Όπως είπε η Επίτροπος, η διαφορά ή έγκυται στο γεωγραφικό προσδιαρισμό μιλούμε ε, διαφορετικά, αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή και τη διάσταση των φύλων διαφορετικά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και βεβαίω θέλουμε να γίνεται gender mainstreaming και να συμπεριλαμβάνονται τα θέματα του φύλου στη χάραξη πολιτική για την κλιματική αλλαγή. Και η Επίτροπο πήρε το λόγο προηγουμένω, παρουσίασε διάφορα παραδείγματα. Υπόθηκε ότι οι γυναίκε είναι πιο εκτεθειμένε στα πλήγματα τη κλιματική αλλαγή και προσαρμόζονται κιόλας. Θα πρέπει να πετύχουμε ισότητα των φύλων όταν γίνεται λόγος για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Μιλήσαμε για το Παγκλατές, για τους εκτοπισμένους λόγω πλημμυρών το ίδιο και στο Βιετνάμ. Ακούσαμε πολλά τέτοια ε, παραδείγματα σήμερα και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ευπάθεια, με την ευαισθησία, με την ε, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με τη μείωση της εκπομπής ε, αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ούτω καθεξής. Πλήττονται οι γυναίκες περισσότερο για πάρα πολλούς λόγους και πολύ γνωστούς λόγους. Επομένως, σε ό,τι έχει να κάνει με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην πολιτική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, εκεί σε αυτό το πεδίο ε, δρούμε περισσότερο και συμπεριλαμβάνουμε τη διάσταση του φύλου σε αυτού του είδους την πολιτική, σε αυτό το σκέλος δηλαδή της πολιτικής της κλιματικής αλλαγής, το σκέλος που έχει να κάνει με την προσαρμογή. Υπόθηκε ότι η διάσταση του φύλου θα πρέπει να ενταχθεί σε όλες τις πολιτικές που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Εγώ θέλω να εστιάσω περισσότερο στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για τους λόγους που σας εξήγησα και στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει ένα νέο φάκελο, αν θέλετε, στο χαρτοφυλάκιό μας. Έχουμε 20 χρόνια νομοθεσίας για τα θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Έχουμε ε, πάρα πολλά ε, νομοθετήματα. Θα μπούμε στη τρίτη φάση ε, του συστήματος εκπομπής ρήπων. Ωστόσο, το 2007 ξεκινήσαμε με την πράσινη βίβλο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή πράσινη βίβλος η οποία προέκυψε μετά από αίτημα μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία οι μέλη ζητούσαν να μάθουν πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό το θέμα ή όχι και μετά τη διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη και τους ενδιαφερόμενους φορείς και με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο στήριζε εμάς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθειά μας και εκτιμούμε ιδιαίτερο τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν μετά από όλα αυτά το 2009 δημοσιεύσαμε τη Λευκή Βίβλο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και εκεί παρουσιάζουμε κάποιους πυλώνες όπου... Ε, ε, πάνω στους οποίους θα στηρίξουμε τα πιο σημαντικά ζητήματα. Επομένως, η διάσταση των δύο φύλων είναι ένας από αυτούς τους πυλώνες, αν θέλετε, η ανάπτυξη μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση, ε, συμπερίληψη της κλιματικής αλλαγής στις υπόλοιπες πολιτικές, ρόλος των ε, εργαλείων της αγοράς όπως είναι η ασφάλιση και το καθεξής. Αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες και στηρίζονται σε πολλά θεμέλια. Ένα θεμέλιο από αυτά είναι και η διάσταση των δύο φύλων. Όταν λοιπόν ε, συγκροτήσαμε την ομάδα εμπλεκόμενων φορέων ε, και είχαμε και το, την ομάδα καθοδήγησης τον ε, περασμένο Σεπτέμβριο είχαμε δώσει καταπευθυντήρες γραμμές ε, για την διάσταση των δύο φύλων και όταν προσαρμόσαμε τη στρατηγική για το 2013 η οποία θα είναι και η συνέχεια της ε, Λευκής Βίβλου του 9 και της ανακοίνωσης του 2007 τότε συμπεριλάβαμε και πάλι αυτή τη διάσταση των δύο φύλων. Τα λέω όλα αυτά συνοπτικά και εντάχει για να σας πω ότι ε, σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή έχουμε συμπεριλάβει όπου μπορούμε τη διάσταση του φύλου. Σε θέματα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής ε, και το πόσο μπαίνει εκεί μέσα η διάσταση του φύλου, σε αυτά δεν θα επεκταθώ γιατί η Επίτροπος τα ανέφερε επανειλημμένος. Από εκεί και πέρα Όντω ε, θα πρέπει οι γυναίκες να συμμετέχουν περισσότερο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ε, που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό το επιτυχάνουμε μέσω της ομάδας των εμπλεκόμενων φορέων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τρεις θέσεις σε αυτή την ομάδα και εκπροσωπείται. Ο κύριος Πρόντι είναι επίτιμο μέλος και είναι πάντοτε παρόν. Στις 8 Νοεμβρίου θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση της ομάδας αυτής. Και θα ήθελα τέλος να κάνω μία-δύο παρατηρήσεις σε σχέση ε, με τις ομιλήτριες. Ε, να ξεκινήσω από την παρέμβαση που είχε να κάνει με τη χρηματοδότηση των πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Βάσει του UNFCCC και βάσει της συμφωνίας της Κανκούν λαμβάνεται πλέον υπόψη το θέμα της ισότητας των φύλων ε, στις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή και σε όλες τις δράσεις και τις πολιτικές. Τώρα για τα οικονομικά ζητήματα στα οποία αναφερθήκατε και είπατε ότι θα πρέπει να τα παρακολουθούμε ο πράγματι σε σχέση με τη χρηματοδότηση Fast Start η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διατηρήσει τις δεσμεύσεις της 100 δις ευρώ ε, το χρόνο μέχρι το 2020 και θέλουμε πάντοτε να στοχεύουμε τις πιο ευπαθείς ή τις πιο φτωχές ομάδες, τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τις ε, πιο φτωχές χώρες οι οποίες είναι και νησιωτικές. η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει τις δεσμεύσεις της και τη στηρεί. Ε, αθρηστικά έχουμε 2,4 δις ευρώ, δηλαδή το 1 τρίτο αυτού που συλλογικά έχουν υποσχεθεί και δεσμευθεί οι ανεπτυγμένες χώρες. Και 200 εκατομμύρια ευρώ ε, από το 2009 μέχρι το 2010 ε, θα διοχετευθούν μέσω της Συμμαχίας για την Κλιματική Αλλαγή. Βλέπετε λοιπόν ότι είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητές, το είπατε κι εσείς και να σας πω ότι για το fast start ε, χρηματοδότηση αυτή και για τις μακροπρόθεσμες δεμεύσεις δεν έχουμε ξεφύγει, ε, ούτε έχουμε καθυστερήσει στην εκταμείευση των κονδυλίων που έχουμε υποσχεθεί και που έχουμε δεσμεύσει για τέτοιου είδους δράσεις. Και τέλος. Υπήρξαν αιτήματα για πιο φιλόδοξες διαπραγματεύσεις βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Όσο περισσότερο μειώσουμε τις εκπομπές ρήπων, τόσο λιγότεροι θα κληθούν να προσαρμοστούν και να, θα αναγκαστούν να πληγούν. Και γι' αυτό θέλω να σας πω ότι η Ευρώπη ήταν η πρώτη ε, Ήπειρος και ο πρώτος οργανισμός που υιοθέτησε τέτοιου είδους νομοθεσία, μείωση κατά 20% μέχρι το 2020 κτλ. Εμείς ε, ε, είμαστε σε φάση επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί με το πρωτόκολλο του Κιώτο δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας, ούτε μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μόνοι μας, αν δεν μας ακολουθήσουν οι ΙΠΑ και οι αναδυόμενες οικοδομίες. Θα πρέπει και αυτές να κάνουν ε, το μάτι που τους αναλογείς και ε, ζητούμε και την Ευρωπα... τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να πείσουμε όσους δεν έχουν ακόμα πιστεί έξω από την Ευρωπαϊκή Επικράτεια ότι πλέον έχει έρθει η ώρα να αλλάξουμε τις συνήθειες και για να αλλάξουμε και την κοινωνία μας. Θέλετε να απαντήσετε ναι. Θα ήθελα εν συντομία να σχολιάσω το θέμα της χρηματοδότησης της ε, κλιματικής πολιτικής, να επισημάνω το θέμα της ποσότητας αλλά και της, ποσ... της ποιότητας της κλιματικής χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, περισσότερα κονδύλια διοχετεύθηκαν προς το μετριασμό ε, παρά προς την προσαρμογή. Και αυτό πλήττει τα δύο φύλλα διαφορετικά. Άρα ε, οξύνει τη διάσταση του φύλου. Και επίσης η Ευρώπη ενίοτε δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Δηλαδή κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιεί το δικό της ορισμό και βασίζεται σε δικές της γραμμές βάσης. Όντως γενικώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ξεφύγει από, τα, από τις δεσμεύσεις της, ε, τηρεί τις δεσμεύσεις της, αλλά μπορεί να κάνει περισσότερο για να χρηματοδοτηθεί περισσότερο το σκέλος της προσαρμογής σε σχέση με το σκέλος του μετριασμού, προκειμένου να καλυφθεί ε, απόσταση, ε, η οποία παραμένει αυτή τη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά την Παγκόσμια Συμμαχία για την Αλλαγή του Κλίματος, το GCCA, δεν είμαι εμπειρογνώμων φυσικά ούτε ειδική, απλά να σας πω ότι έχω διαβάσει. Ε, δίνεται εκεί προσοχή σε κάποια σημεία που τονίζουν τη σχέση με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τις πιο φτωχές. Μείωση ε, των εκπομπών ρήπων λόγω της ε, Αποψήλωση των δασών π.χ. Είναι πράγματα αυτά που αφορούν πάρα πολύ τις ε, γυναίκες. Στη διαδικτυακή τοποθεσία της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Κλιματική Αλλαγή δεν γίνεται καμία αναφορά στα θέματα των δύο φύλων και είδα και την ανακοίνωση του 2007. Εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει μόνο μία φορά τις γυναίκες ως μία από τις ε, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Και ένα θέμα είναι να αναγνωρίζει κανείς το ευπαθές της των γυναικών, αλλά δεν αρκεί να παραμένει κανείς μόνο σε αυτό. Το ε, πλαίσιο εφαρμογής της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την κλιματική αλλαγή, αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί όπου προσδιορίζεται ο τρόπος υλοποίησης. Ε, λοιπόν, εκεί δεν γίνεται αναφορά στις γυναίκες ή στα ανθρώπινα δικαιώματα και το καθεξής. Δηλαδή, το λέω για να πάντοτε να, να μην ξεχνούμε να συμπεριλαμβάνουμε αυτού του είδους τις παραπομπές και τις ε, διατυπώσεις σε όποιο κείμενο ε, και αν έχουμε ή σε όποια πολιτική και αν χαράσουμε ή υλοποιούμε. Ευχαριστώ η Ροσάριο Μπέντο Παΐς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, για την ποιότητα της χρηματοδότησης, για τις δράσεις κλίματος, να σας πω καταρχάς ότι μπορώ να μιλήσω μόνο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή είναι εκπροσωπώ εδώ. Δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά ή της, ε, ε, γιατί υπάρχουν θέματα επικουρικότητας και εθνικής ε, κυριαρχίας ως προς την χρηματοδότηση. Υπάρχει ένα σκέλος το οποίο το αποφασίζουν τα κράτη-μέλη μόνο. Το Fast Start Financing, η χρηματοδότηση αυτή, αφιερώνει 5% των κονδυλίων στον μετριασμό και 5% στην ε, προσαρμογή. Και ε, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλα τα ε, καινούργια προγράμματα ε, έχουν νομίζω επιπρόσθετη αξία. Ε, βέβαια μπορούν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να σας απαντήσουν με πιο πολλές λεπτομέρειε για το τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο και στην εκλογική τους περιφέρεια. Τώρα, στο, ως την Παγκόσμια Συμμαχία για την Κλιματική Αλλαγή, θα το αναφέρω αυτό στους συναδέλφους, αυτό το οποίο είπατε, αλλά να σα πω ότι αυτή η συμμαχία είναι για τι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε, τι νησιωτικέ και τι πιο φτωχέ. Και βεβαίω η συμμαχία αυτή θέλει να βοηθήσει τι πιο ευπαθείς ομάδε ενό κοινωνικού συνόλου. Και βεβαίω οι γυναίκε είναι μεγάλο μέρο αυτή τη ε, ευπαθούς ομάδα και άρα τη αφορά η χρηματοδότηση αυτή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, είναι μια πρωτοβουλία μόνο για τις νησιωτικές και λιγότερο ανεπτυγμένες μικρές χώρες. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι γυναίκες σε αυτές τις χώρες πλήττονται περισσότερο, όντως. Θα, το, το λοιπόν και θα το μεταφέρω στους αρμοδίους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Καλώς, λέει ο Πρόεδρος. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια από ό,τι βλέπω. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, θέσω αυτό το ερώτημα. Έχετε σχόλια, έχετε παρατηρήσεις, έχει έρθει τώρα η ώρα να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ. Και να δηλώνετε το όνομα και την ιδιότητά σας. Λέγομαι Χάτσνικ και είμαι μέλος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Φλόρα. Είμαστε ένα δίκτυο ειδικών για την ε, για, το, για τα δύο φύλλα, την αηφορία και το οικονομικό αυτό σκέλος. Μία γενικότερη ερώτηση για το σύνολο της συζήτησης. Η κλιματική αλλαγή είναι το αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου μοντέλου οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης. Μήπως τελικά αυτό το μοντέλο οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης είναι αυτό που προκαλεί ε, την κλιματική αλλαγή και ε, λειτουργεί τελικά ως ένα ποτάμι το οποίο ρέει, ποτάμι επιπτώσεων και καθόλου τη διάρκεια της ροής του ποταμού βλέπουμε ότι οι γυναίκες βρίσκονται ε, στο ε, τελικό στάδιο εκεί που ο ποταμός χύνεται στη θάλασσα για να το πω μεταφορικά και άρα γι' αυτό πλήττονται και περισσότερο. Και ένα ερώτημα προς την κυρία Πιετικάινεν. είναι έχει γίνει μια ανάλυση της ε, διάστασης των φύλων ως προς την επιλογή μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης. Οι γυναίκες δεν συμμετέχουν στη διαμόρφωση αυτού του οικονομικού μοντέλου και έτσι δεν έχουν ε, θέσεις όταν ε, διατυπώνονται προτάσεις για λύση των προβλημάτων. Θα ήθελα να προτείνω, και αυτό ουσιαστικά απασχολεί την μη κυβερνητική οργάνωση, στην οποία εργάζομαι να προβλέψουμε ακριβώς τέτοιου είδους ε, δράσεις. Όχι μόνο στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, αλλά και σε άλλες δομές, πολιτικές ή οικονομικές, το πρόβλημα είναι πάντοτε ίδιο και παντού. Δηλαδή είναι δομικό το πρόβλημα και χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές για την αλλαγή αυτού του μοντέλου του ευρύτερου. Ε, δεν δεν ξέρω σε ποιον θα πρέπει συγκεκριμένα να απευθύνω το ερώτημα. Ερωτώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να ασχοληθεί με την πηγή του προβλήματος, από πού πηγάζει το περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα που οδηγεί μεταξύ άλλων και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και στην υποβάθμιση του ρόλου της γυναίκας. Ευχαριστώ. Δεν είμαι σίγουρος ποιος θα μπορούσε να απαντήσει το ερώτημα αυτό. Δεν ξέρω αν θέλει κι άλλο το λόγο. Εγώ έχω σπουδάσει οικονομικά και γνωρίζω πολύ καλά τη συζήτηση αυτή. Όντως γίνεται η συζήτηση για το πώς μπορεί κανείς να δομήσει αυτή την ε, ιδέα της οικονομίας και πώς μπορεί να υποφεληθεί τι περιλαμβάνει η ευημερία, ποιο είναι το κόστος και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Εγώ είμαι υπέρ του να γίνονται τέτοιες τέτοιες συζητήσεις. Βεβαίως μετά είναι ένα άλλο θέμα το αν θα μπορούσαμε να υποφεληθούμε καλύτερα μέσω μιας άλλης προσέγγισης αυτήν την έκθεση. Ε, δεν ξέρω η συγγύτρια ίσως θα μπορούσε να απαντήσει καλύτερα για το πώς δηλαδή διαχειριστήκαμε τα οικονομικά μοντέλα. Please. Άλλος κανείς, παρακαλώ. Ευχαριστώ για το σχόλιο. Όντως είναι σημαντικό να δούμε ποια είναι η πηγή όλων αυτών των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Και νομίζω ότι υπάρχει και μεγάλη, μια μεγάλη ευκαιρία στις συζητήσεις του Ρίο 20 για τις ε, πράσινες οικονομίες. Ποια δηλαδή οικονομία είναι αυτή που θέλουμε και ποια κοινωνία τελικά είναι αυτή που θέλουμε. Υπάρχει και μια πιο ολιστική προσέγγιση η οποία χρειάζεται αλλά λείπει γιατί ακόμα έχουμε προσανατολιστεί κυρίως στα τεχνολογικά στοιχεία της υπόθεσης. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να προσθέσω απλώς για την πράσινη οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ανακάλυψα ότι δεν υπάρχει ε, gender mainstreaming στο σημείο αυτό. 8% των ε, θέσεων εργασίας στην πράσινη ανάπτυξη, στην πράσινη οικονομία καλύπτονται από άντρες. Το 80% των ε, θέσεων εργασίας καλύπτονται από άντρες. Δεν θα πρέπει λοιπόν να προωθούμε επενδύσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίς να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν και θέσεις για γυναίκες. γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να απαλείψουμε αυτή την, αυτό το μεγάλο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Μάλιστα, χτες η Δανία εξέδωσε μία έκθεση από τα συνδικάτα που λέει ότι τα νεαρά κορίτσια που δουλεύουν σε θέσεις εργασίας στον τομέα των κατασκευών δεν μπορούν να κάνουν μια μαθητεία γιατί τους αρνούνται την, τη θέση. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Πρέπει να δούμε το θέμα των γυναικών και των πράσινων θέσεων εργασίας. Εγώ συναντήθηκα στη Βραζιλία, στο Σαο Παόλο, με συνδικαλιστές και μου είπανε ότι έχουν πολλά προγράμματα μαζί με χώρες όπως η Γερμανία, η Ισπανία και άλλες για αυτό ακριβώς το θέμα, γυναίκες και πράσινες θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το δούμε όταν μιλούμε για την οικονομία και για την πράσινη οικονομία. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάιναν. Σύντομα να το πω για να το λάβει υπόψη της η εισηγήτρια. Στα οικονομικά υπάρχουν δύο βασικές ε, σκέψεις, ότι υπάρχει μια τελείωτη ε, ανάπτυξη χωρίς όρια, ότι δηλαδή δεν θα υπάρχουν όρια για τίποτα και υπάρχει και μια άλλη σκέψη που βασίζεται στην κυκλική τύχη της ε, οικονομίας και στους πόρους της και στο, στους περιορισμούς που τελικά υπάρχουν. Αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά δεδομένο και θα μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε. Το δεύτερο δηλαδή, τη δεύτερη πτυχή, θα μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε στην έκθεση για την αποδοτικότητα των πόρων, για το, για το κόστος. Ίσως θα μπορούσαμε να το βάλουμε και στον οδικό χάρτη που προέκυψε από την Κομισιόν συνδέοντας έτσι και το όλο θέμα με τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Δεν βλέπω άλλον κανέναν να ζητάει το λόγο. Ωραία. Οπότε να δώσω το λόγο στην κυρία Νίλσεν για τα καταληκτικά σχόλια. D'abord, je vous remercie. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ε, ευχαριστήσω όλους και όλες για τα όσα μας είπαν και θα μας, που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην εκπόνηση εκθέσεως ε, με θέματα αυτά. Για όσους δεν ήταν εδώ πριν, ότι, να πω λοιπόν ότι η Επίτροπος αναφέρθηκε προηγουμένως ε, στο θέμα των γυναικών στα πλαίσια της πράσινης οικονομίας. Ε, και άλλωστε πρόκειται, έναν, ε, πρόκειται για έναν από τους στόχους τους οποίους θέλουμε να επιτύχουμε. Εν συμπεράσμετη θα ήθελα να πω ότι το διακύβευμα, η πρόκληση του αιώνα είναι βεβαίως ο αγώνας κατά της ε, κλιματικής αλλαγής και η μεγάλη αυτή πρόκληση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τη συμμετοχή του άλλου μισού του ουρανού τις γυναίκες δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό είναι προφανές. Ε, αυτή η πρόκληση είναι ε, μίζωνος σημασίας και είμαι απολύτως πεπισμένη ότι χωρίς ε, τη συμμετοχή του μισού και παραπάνω του πλανήτη, τότε θα ασφαλώς στην καταστροφή. Εάν θέλουμε να σώσουμε αντιθέτως τον πλανήτη, θα πρέπει με κάθε τρόπο να συμμετάσχουν οι γυναίκες οι οποίες βεβαίως συμφωνώ δεν είναι μονάχα θύματα, έστω και αν διαπιστώνουμε ότι συχνά, υπερβολικά συχνά μάλλον, σε φυσικές καταστροφές οι γυναίκες ε, είναι τα πρώτα και περισσότερα θύματα. Αλλά όπως λαμπρά μας έχει καταδείξει ο Αγκαρή Ματάη και άλλες ε, γυναίκες υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες σε συνειδητοποίησαν τα πράγματα, πήραν τα πράγματα στα χέρια τους, συνειδητοποίησαν την δύναμή τους και έχουν ήδη επιφέρει λύσεις. Τι μας βαθαίνουν αυτές οι γυναίκες, ότι όταν λαμβάνονται υπόψη οι γυναίκες τότε διευρύνεται το πεδίο σκέψης μας. Και με τα παραδείγματα που έδωσε και προηγουμένω, κατέστησε σαφέ ότι κάθε φορά που λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των γυναικών, τότε ε, υποβάλλονται νέε λύσει, προβάλλονται νέε σκέψει και τελικά συνειδητοποιούμε ε, ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος. Πρέπει να πω επίσης ότι υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι η απόλυτη προτεραιότητα είναι η κλιματική αλλαγή και μετά ακολουθούν ε, τα ε, δικαιώματα των γυναικών. Ξέρουμε αυτούς που ορθώνουν αυτόν τον λόγο και ξέρουμε ότι ιστορικά έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η αντιμετώπιση. Ας κάνουμε πρώτα την, ε, ας κάνουμε πρώτα την επανάσταση και θα λύσουμε το θέμα των γυναικών μετά. Όχι. Όχι. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά. Δεν είναι δυνατόν να ε, ε, ε, αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις χωρίς να λάβουμε υπόψη μας από την πρώτη στιγμή της γυναίκες. Η ανθρωπότητα, λέω, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα σημαντικά παρά μόνο με συμμαχία όλων των ανθρωπίνων δυνάμεών της. Στην Αφρική οι γυναίκες συμμετέχουν κατά 83% στην παραγωγή τροφής. Γι' αυτό οι Αφρικανές γυναίκες ξέρουν περί πρόκειται, συνειδητοποιούν την προβληματική και δεν είναι τυχαίο. Ε, ξέρουν, γνωρίζουν, αυτές διαχειρίζονται τη γεωργία ε, και αυτές διαχειρίζονται τα θέματα διατροφής Επομένως λέγω ότι λαμβάνοντα υπόψη τις γυναίκες, τις ανάγκες τους, τις ε, διεκδικήσεις τους, ε, τις επιθυμίες τους, ε, αυτό δεν αποτελεί πρόσκομα στις διαδικασίες, αλλά ευκαιρία. Μια ευκαιρία μετάδοσης των παραδοσιακών πατρογονικών γνώσεων, μια ευκαιρία να αλλάξουν οι κατανολικές συνήθειες, μια ευκαιρία να βρεθούν τοπικές συγκεκριμένες λύσεις. Τελικά μια ευκαιρία για να ε, ξεπεραστούν οι πιο ε, γνωστές ε, διακρίσεις, αυτές δηλαδή οι οποίες βασίζονται στο φύλλο. Φυσικά μακριά από μας οι έτοιμες λύσεις και οι απλοϊκές αντιμετωπίσεις. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει ταυτοχρόνως να κινηθούμε έτσι ώστε να αυξήσουμε την αντιπροσωπευτικότητα των γυναικών σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι θεμελιώδου σημασία. και πρέπει οπωσδήποτε να επιτύχουμε αύξηση της αντιπροσωπευτικότητας των γυναικών. Ε, θέλουμε ισότιμη παρουσία των γυναικών σε όλα τα θεσμικά όργανα. Δεύτερον, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε την δυνατότητα να δράσουμε με τρόπο ευφύ ε, να έχουμε συνολικά στοιχεία όπως αναφέρθηκε από την προηγούμενη ομιλήτρια ε, και συστηματικά να έχουμε στοιχεία αναφύλο Οποτεδήποτε ξεκινάει ένα πρόγραμμα, οποτεδήποτε εκπονείται μια στρατηγική, να γίνεται η προσπάθεια να συμμετέχουν οι γυναίκες στις διαπραγματεύσεις, στις διαβουλεύσεις και ε, ε, στον προγραμματισμό των δράσεων και ως ε, μέλος ε, της Επιτροπής ε, Δικαιωμάτων των Γυναικών πραγματικά πιστεύω ότι αυτά είναι πολύ βασικά πράγματα και πρέπει να αγωνιστούμε έτσι ώστε να τα επιτύχουμε. Δώσαμε προηγουμένως συγκεκριμένα παραδείγματα, έδωσα και εγώ. Δεν χρειάζεται να επανέλθουμε, όμως Ε, πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο τα πράγματα και να διευρύνουμε τη σκέψη μας όσον αφορά ε, την ε, ε, κλιματική αλλαγή. Να τελειώσω λέγοντας ότι η συμπερίληψη ε, των γυναικών στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών οπωσδήποτε δεν είναι πρόσκομα, αλλά ε, θα διευκολύνει τον αντίον την αντιμετώπιση του προβλήματος με τρόπο γρηγορότερο και αποτελεσματικότερο. Θα πρέπει επομένως να δράσουμε ε, σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, σε επίπεδο κρατών μελών, παντού. Πριν τελειώσω θα ήθελα να σας διαβάσω την ε, φράση που είπε η κυρία Μασαμπανέ, Υπουργός Εξωτερικών ε, της ενότητας Αφρικής, η οποία θα προεδρεύσει ε, την διάσκεψη COP17 στο Ντέρμπαν. Λέει λοιπόν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να χειροκροτούμε μονάχα με ένα χέρι ή να περπατάμε με ένα μόνο πόδι. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι σαφές και δείχνει πώς βλέπουμε τα πράγματα. Να πω επίσης ότι όσοι ενδιαφέρονται για την ε, ε, συνέχιση της συζήτησης αυτής να πω ότι αύριο οργανώνεται σε Βρυξέλλες σε ένα εργαστήρι, ένα workshop ε, και η γραμματεία μπορεί να σας δώσει πληροφορίες. Εάν μερικοί ή μερικές μεταξύ ημών επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό το εργαστήρι σας λέγω ότι θα έχουμε την δυνατότητα ε, εμβάθυνσης ε, με τις πανελίστριες ε, των θεμάτων αυτών. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σύντομα. Det här är väldigt spännande. Ε, Πιστεύω ότι τα ζητήματα τα οποία συζητήσαμε σήμερα, αυτή, αυτό το πράσινο όραμα μας αφορά όλους και όλες. Ε, όσον αφορά τον τρόπο ζωής, ναι, ήθελα να πω ότι πραγματικά πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Αλήθεια είναι αυτό. Επίσης αληθεύει ότι οι άνδρες δυσκολεύονται περισσότερο στο να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους ενώ μια γυναίκα πιο εύκολα αποφασίζει να αλλάξει τη ζωή της. Μερικοί νομίζουν ότι το να αλλάξουν κάποια συνήθεια στη ζωή τους σημαίνει μια έλλειψη, σημαίνει μια στέρηση. Δεν είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, αν στο κοινοβούλιο μας λέγανε πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις τις συνεδριάσεις και να μειώσει συνεδριάσει κατά 50%, ε, ε, εγώ θα το έκανα. Θα το έκανα. Και θα είχα την εντύπωση, όχι απαραίτητα ότι βελτιώνω ε, την ποιότητα ζωής μου, αυτό είναι κάτι διαφορετικό, αλλά θα μπορούσαμε να μειώσουμε, ας πούμε, άνετα τις συνεδριάσεις ser stor betydelse av att det finns i de enskilda länderna. Είναι αλήθεια όλα αυτά που ακούσαμε. Είναι αλήθεια επίσης ότι υπάρχει δέσμευση σε πολλές χώρες, σε τοπικό επίπεδο. Στο, επίπεδο της ε, κοινωνίας, έτσι ώστε να αναλυθούν κοινέ δράσεις. Ε, επίσης ε, υπάρχουν χώρες που έχουν ήδη ξεκινήσει να αλλάζουν ε, την, ε, τον τρόπο σκέψης και να συμπεριλαμβάνουν τις γυναίκες στην χάραξη στρατηγικής, ε, στις συγκοινωνίες, στις, οπουδήποτε. Οι γυναίκες σαφώς δεν είναι μόνο θύματα, σαφέστατα μπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην πολιτική περιβάλλοντος ε, μπορούν να ληφθούν, να αναλυφθούν συγγνώμη δράσεις οι οποίες θα βασίζονται ε, στην ισότητα των φύλων. Αυτά τα λίγα είχα να πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δώσατε και τις οποίες βεβαίως θα λάβουμε υπόψη μας ε, στην μελλοντική μας εργασία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις τέσσερις κοιόδες εισηγήτριες και φυσικά την κυρία Κιλ που είναι και η συγγήτρια. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη γνωμοδότησή σας. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης εξεπροσωπήθηκε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και την ε, γραμματεία η οποία διοργάνωσε ε, και κατέστη, διοργάνωσε αυτήν την ε, ακρόαση. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να την κάνουμε. Θα ήθελα τελικώς να ευχαριστήσω και κυρίως να ευχαριστήσω όλους τους γερμηνείς για την εξαίρετη εργασία τους. Ευχαριστούμε πολύ και τον Πρόεδρο και οι γερμηνείς τον ευχαριστούν δηλαδή. Ε, ε, οι διερμηνείς μας έδωσαν τη δυνατότητα να εκφραστούμε στις γλώσσες μας. Να ευχαριστήσω τελικά όλους όσους ε, συμμετέσχουν σε αυτήν την ακρόαση. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.